το Ευρωπαϊκού Νοτεξιακού Ταμείου, το ζήτημα των ε, λογαριασμών του ελέγχου των δημοσιονομικών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεσματικότητα στην χρήση των δαπανών του Ευρωπαϊκού προπολογισμού όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και βεβαίω την καταπολέμηση των απατών. Είναι ευρύτατο το χαρτοφυλάκιο. Έχουμε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καλή συνεργασία σε όλα αυτά τα θέματα που έθιξα. Θέλουμε να προχωρήσουμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε σε καλή συνεργασία σε όλα αυτά. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια καλή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. 25 ήταν οι πρώτε ερωτήσει που κατέθεσε προκαταβολικά αυτή τη συζήτηση η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σα ευχαριστούμε πολύ για τι απαντήσει και βεβαίω θα επανέλθουν οι συνάδελφοι με επιπλέον πρόσθεσε ερωτήσει και παραδίδω πάλι το λόγο στον Πρόεδρο. Ευχαριστούμε και το λόγο ο Παύλ Ζόμπεντα, ο Πρόεδρο τη ε, Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω από πλευράς της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ότι με μεγάλη μας χαρά έχουμε εδώ τον Επίτροπο Έτιγκερ. Γνωρίζετε αγαπητέ Επίτροπο ότι το νέο σας χαρτοφυλάκιο θα καλύψει και τους ανθρωπίνους πόρους και όπως αναφέρεται επιλέξει συνορισμός του προσωπικού και της Διοικητικής Επιτροπής, το, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, προσλήψεις, ε, κινητικότητα προσωπικού και επίσης θα εξασφαλίσετε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και άλλα. Ε, η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, είναι αρμοδία μεταξύ άλλων, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική, να είναι αμερόληπτη η δίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, αυτά προβλέπονται στο 298 και το 96 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, η Νομική Επιτροπή ανυπόμενα περιμένει να τα συζητήσουμε τα σχετικά απόψε και θέλουμε ότι θα είναι πάρα πολύ παραγωγική η συζήτησή μας. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, εμείς λέει ο πρόεδρος και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος Έτιγκερ για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε Ορτσβή, Κυρία Πρόεδρε Γκρέστιλε, αγαπητέ κύριε Σφόποτα, κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καταρχάς μια πολύ καλή χρονιά για σας προσωπικά, επαγγελματικά, σε εσά και τους συνεργάτες σας, να είναι επιτυχές το 2017. Το Κοινοβούλιο οργανώσει μια ε, ακρόαση πριν από δύο χρόνια για την υποψηφιότητά μου ως Επιτρόπου Αρμοδίου για τα θέματα της ψηφιακής οικονομίας και πολλά από αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει έχουν προχωρήσει υπό τη δική μου καθοδήγηση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο το 2017 μαζί με το Συμβούλιο θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση κρίσιμων προστάσεων και ε, συζητήσεις. Και τώρα έχουμε το θέμα του προϋπολογισμού και του προσωπικού. Με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα μελετώ τις προτάσεις σας και τις ε, ιδέες σας. Ήθελα να επισημάνω πως ανέκαθεν με ενδιέφερα τα θέματα του προϋπολογισμού και του προσωπικού. Είμαι δικηγόρος, επί 26 χρόνια βουλευτής ε, του, της Βάδης Βιτεμβέργης, περιφέρειας Ευρώπης, επί 5 χρόνια επικεφαλής τοπικής κυβέρνησης, με προϋπολογισμό της Βάδης Βιδεμβέργης περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, με θέματα που έφταν, με ποσά που έφταναν περί, τα, περί τους 230.000 εργαζομένους περιλαμβανομένων και των, και των ε, αστυνομικών και λοιπόν δυνάμεων. Είχα εντωμεταξύ στις αρμοδιότητες μου ως Επιτρόπου την δυνατότητα να ασχοληθώ με την ψηφιακή Ευρώπη, με την ε, κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια ε, και επικοινωνίες και μπόρεσα πιστεύω να συμβάλλω στην δουλειά της προηγούμενης, των προηγουμένων επιτρόπων στον προπολογισμό του κ. Λεβαντόφσκη αλλά και της κυρίας Γεωργίευα. Έχω μια κάποια λοιπόν εμπειρία να προσφέρω από την προηγούμενη μου εργασία. Αλλά έχουμε εδώ παρόντες τους τρεις προέδρους των επιτροπών και γνωρίζω ότι και οι τρεις επιτροπές είναι συναρμόδιες. Εδώ εγώ έχω να προσφέρω τη βούλησή μου για έναν διαφανή, ουσιαστικό διάλογο για τα επόμενα χρόνια, για αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προπολογισμό, για μια ευφυή πολιτική για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός είναι ένα από τα κύρια ε, δικαία των δημοκρατιών από τις πιο παλές, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις και τις πιο νέες και γι' αυτό αναγνωρίζω το ενδιαφέρον το που έχετε αλλά και τις μεγάλες φιλοδοξίες για έναν προπολογισμό ο οποίος θα υπηρετεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία σχετική με τον προπολογισμό και την εκτέλεσή του είναι ε, αρμοδιότητες που και το Κοινοβούλιο από με το Συμβούλιο, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις εθνικές, τις περιφερειακές αλλά και τις τοπικές ένωμες τάξεις. Έχουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή κουλτούρα της άσκησης ε, του δημοσιονομικού δικαίου ε, που συνεχίζεται και διατηρείται. Για το προσωπικό. Έχουμε να κάνουμε με προσωπικό ύψης της ποιότητας, κίνητρα λοιπόν, εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες και περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού μας πρέπει να είναι κύριοι στόχοι μας. Χρειάζεται να έχουμε τα καλύτερα μυαλά, τα πιο ευφυή μυαλά στα θεσμικά μας όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, σε όλα τα όργανα και βέβαια πάνω απ' όλα στην Επιτροπή. Έχουμε καλούς υπαλλήλου, άντρες και γυναίκες και έχουμε και την ευκαιρία πιστεύω να προσελκύσουμε τους ικανότερους από τα κράτη-μέλη. Πρέπει ταυτόχρονα όμως να έχουμε υπόψη και τις συνθήκες ε, οι οποίες επικρατούν στην, στην ιδιωτική αγορά και δεν πρέπει έναντι αυτής, αυτών των δυνατοτήτων εμείς να υπολοιπόμεθα έτσι ώστε να προσφέρουμε καλές ευκαιρίες απασχόλησης για το προσωπικό μας. Χρειαζόμαστε μια δραστήρια πολιτική για το προσωπικό. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η κινητικότητα του προσωπικού μας, η δυνατότητα για περαιτέρω κατάρτιση και ιδιαίτερος βεβαίως Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο 40% των ε, θέσεων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όπως προβλέπονται για το, για το τέλος του 2019. Πρέπει να επιτύχουμε το ποσοστό αυτό. Ε, θα δείτε βεβαίως ότι στη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια αλλά και για τη Γενική Διεύθυνση ε, Ψηφιακής Οικονομίας είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να επιτύχω σημαντικές εξελίξεις για την ανάπτυξη αυτών των θέσεων στελεχών. Η πολυπικιλότητα, η ανοιχτή συμμετοχή, η ισότητα ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους, η απουσία διακριτικής μεταχείρισης είναι δεσμεύσεις τις οποίες έχω να λάβει και εξακολουθώ να ε, διατηρώ. Ιδιαίτερα λοιπόν για ομάδες προσωπικού που μπορεί να έχουν μια ιδιαιτερότητα όπως η ΛΟΑΔΜ αλλά και άλλε πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα δικιά τους και να ακούγονται οι διεκδικήσει τους. Έχουμε σε σχέση με τον προπολογισμό για το προσωπικό μας περί το 6% έλλειμμα σε σχέση με τις ανάγκες μας. Ωστόσο στον τομέα του προσωπικού μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίσουμε ε, εξοικονομήσεις δαπανών με πολύ καλύτερη απόδοση της δουλειάς του προσωπικού μας. Είναι μια προσπάθεια την οποία θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι με ένα ετήσιο ποσοστό του 1% στις περικοπές θα μπορούσαμε να έχουμε 5% περιορισμό των δαπανών και βελτίωσε ταυτόχρονα δομική του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Όπω είπα όμω θα πρέπει και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού μας και της δουλειά του να διαφυλαχθούν. Ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτών βεβαίω θα είναι το ζήτημα του Brexit. Την ειδική αρμοδιότητα έχει στο θέμα αυτό ο πρόεδρος Επιτροπής και ο ε, αρμόδιος εκπρόσωπος του κύριος Μισελ Μπαρνιέ. Ωστόσο και στη δική μου, δική μου τη θέση θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να έχουμε μια καλή, δίκαιη, αποτελεσματική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, τις, ε, για τα ζητήματα που αφορούν τους Βρετανούς υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες και βεβαίω την αντιμετώπιση των ζητημάτων των σχετικών με τη σταξιδότησή του, Μια δίκαιη λοιπόν αλλά και μακροπρόθεσμη συμμετοχή της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τις σχετικέ θαπάνες. Θα είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ σε επικρίσεις που διατύπωσαν τις τελευταίες εβδομάδε κάποιοι εξημών ε, προ το πρόσωπό μου. Θα ήθελα να πω ότι ε, έχω απόλυτη ανεξαρτησία προσωπική από οποιαδήποτε ομάδα πιέσεως ή λόμπι και στα θέματα της ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας είμαι απόλυτο ανεξάρτητος. Ε, μπορώ να ακούσω οποιουσδήποτε έχουν να μου παρουσιάσουν εμπεριστατωμένα στοιχεία με βάση τις ε, προτάσεις τους. Είμαι ως επίτροπος εκείνος ο οποίος είχε περισσότερες συναντήσεις ε, σε σχέση με τα καθήκοντά μου από άλλους συναδέλφους της Επιτροπής. Ιδιαίτερα στον τομέα των, ε, της ψηφιακής οικονομίας έχω να καταδείξω νέες επιχειρήσεις, startups, μικρομεξαίες επιχειρήσεις, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μη ευρωπαϊκές, οι οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο λοιπόν των εργασιών μου έκανα κάθε τι το δυνατό ώστε να έχω συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Είτε ήταν είτε ήταν πολίτης, είτε ήταν εκπρόσωπος της κοινωνίας ή της οικονομίας εκείνος ο οποίος ήθελε να συναντηθεί μαζί μου ε, ο οποίο ήθελε δηλαδή να συναντηθεί με έναν επίτροπο, ήμουν στη διάθεση του κάθε ε, στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου και θα συνεχίσω να το πράττω αυτό. Θα είμαι, σε... θα είμαι λοιπόν να ακούσω, να αφουγκραστώ τον κάθε έναν, αλλά βεβαίω κάθε απόφαση θα ληφθεί με βάση τι προσωπικέ μου εκτιμήσει και τι συμβουλέ που θα μου δίνει το επιτελείο μου. σε σχέση με την ομιλία, κομμάτια της ομιλίας μου στο Αμβούργο πριν από μερικούς μήνες, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν ήταν ούτε είναι πρόθεσή μου να ε, προσβάλλω ή ονδήποτε. Θα ήθελα να εκφράσω ρητά τη λύπη μου για εκείνες τις δηλώσεις, για τον προϋπολογισμό πολύ σύντομα και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο προπολογισμό του 2017 εγκρίνεται και στις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα στηρίξω και τις δικές σας προσπάθειες και βεβαίω ελπίζω ότι και το Συμβούλιο με στι επόμενε ημέρες θα είναι σε θέση να καταλήξει σε μια ε, εφαρμόσιμη πρόταση, σε μια πρακτική πρόταση. Το σημαντικότερο κομμάτι θα το αναπτύξουμε από κοινού με εσάς για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ωστόσο, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και σκοπεύω από το πρώτο εξάμεινο του 2017 προσωπικά να ε, δείξω τη δική μου βούληση για συνεργασία με βάση και την έκθεση Μόντι και τα θέματα των, ε, ιδίων πόρων. Αυτές ήταν οι σύντομε αγωγικέ μου παρατηρήσει και είμαι στη διάθεσή σα για περαιτέρω εμβάθυνση. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε, Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε τους συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε είναι ο πρώτο. Τρία λεπτά για ερώτηση και απάντηση, έτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο, διότι με σαφήνεια παρουσίασε τις προτεραιότητές του. Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευση που αναλαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε για το στόχο που θέτετε, για συνεργασία δηλαδή με το Κοινοβούλιο, για τις μελλοντικές δράσεις, τη μελλοντική συνεργασία και καθ' όλη τη διάρκεια της αδιαδρομής σας ε, φυσικά έχετε καταδείξει την ε, ε, αποτελεσματικότητά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα των πληρωμών, δηλαδή καθυστέρηση των πληρωμών. στο μέτρο που επιστρέφονται 7,5 δις ε, στα κράτη-μέλη και όταν μιλάμε για το Δεκέμβρη του 2016 και έχουμε το 90% των πληρωμών ενώ τον προηγούμενο χρόνο 98% των πληρωμών δηλαδή το 2015 τι πιστεύετε αν προκύψει και πάλι το πρόβλημα των πληρωμών, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξοφλεί τους λογαριασμούς της και θα πρέπει να ε, εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και επειδή τώρα ε, ασχολούμαστε με την αναθεώρηση, αυτό που μας απασχολεί είναι ότι δεν θα καταφέρουμε τελικά να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις μας. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό είκοσι για την απάντηση. Η σημασία των διαρθρωτικών ταμείων για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, και για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για τους νέους. Φυσικά είναι κάτι που δεν μπορούμε να υπερδημίσουμε ενώ φυσικά σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις περιοχές και κυρίως σε χώρες όπως η Πορτογαλία έχουν ιδιαίτερη σημασία και έχουν πλήρη επίγνωση του προβλήματος. Το 2013-2014 υπήρξε πρόβλημα και το έχουμε μελετήσει και μέχρι το 2020 έχουμε προγραμματίσει ε, δράση ε, πολιτικής υποστηρίξης ώστε ε, το 2016 να έχουν ρυθμιστεί τουλάχιστον τα προβλήματα του παρελθόντος. Και θέλουμε να αποφύγουμε στην επόμενη περίοδο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου το ίδιο πρόβλημα. Ε, ε, αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να αποφασίζεται τελευταία στιγμή το τι θα γίνει, όπως το Δεκέμβρη του 2013. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει την υλοποίηση των προγραμματών και τις κατευθυντρίες γραμμές για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Τα κράτη-μέλη θα κάνουν από την πλευρά τους ό,τι μπορούν ούτως ώστε εγκαίρως να κοινοποιούν τα προγράμματα και ταυτόχρονα να έχουμε και μεγαλύτερη ευελιξία, ούτω ώστε από το 2016, 2017 και 2018 όποια κονδύλια δεν έχουν απορροφηθεί να καταστούν διαθέσιμα το 2018-2019, ούτω ώστε να καλύψουμε τα κενά στην καθυστέρηση των πληρωμών. Ευχαριστούμε κυρία Τωμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μεγάλα προβλήματα Παντού υπάρχουν επικρίσεις καθημερινών γιατί παραπονιέται ο κόσμο και δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν, υπάρχει δική, δεν υπάρχει ε, αποτελεσματικότητα. Οπότε θα πρέπει να γίνει κάποιο είδου ανασυγκρότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί τι θεωρείτε, ότι όλα αυτά τα οποία είπατε στο Αμβούργο όσον αφορά τη μετακίνησή σα, ε, αυτό πώ κολλάει σε όλα αυτά. Ε, το τώρα με τι νέε αρμοδιότητε νομίζετε θα ξεχαστούν αυτά Επίσης, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχετε κάθε νομοποίηση στο μέλλον ούτως ώστε να μπορείτε να χειριστείτε και να συζητήσουμε το πολιτές του δημοσιονομικού πλαίσιου του δημοσιονομικού και επίση τι νομίζετε για τι τελευταίε προτάσει του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση του πολιτικού του δημοσιονομικού πλαίσιου. Προτίθεστε να μα υποστηρίξετε έναντι του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Για την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να απεμπλακεί η κατάσταση ε, στο Συμβούλιο με την Μαλτέζικη κυβέρνηση. Έχουμε εντατικότατες επαφές ε, για αυτό το σκοπό. Εάν τελικά στεφθούν με επιτυχία οι προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε να εκπλώσουμε τις προσδοκίες και του Κοινοβουλίου για την επόμενη περίοδο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2020. Θεωρούμε ότι είναι βάσιμα αυτά που ζητάτε και γι' αυτό και ε, επί της αρχής τα υποστηρίζουμε. Ε, τώρα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει συνένεση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Το Συμβούλιο θέλει να χρησιμοποιήσει επίση ε, την αναθεώρηση του πολιτικού του δημοσιονομικού πλαισίου και ενδεχομένω να χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσει πρωτού καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, το πρωί μπορώ να σας δώσω μια ικανοποιητικότερη απάντηση για τον προϋπολογισμό. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ε, θα με διαφάνεια. Θα συνεχίσω να συνεργάζω, να συνεργάζω μαζί σας, να εμβαθύνω ε, τη συνεργασία μας, ώστε να εκπληρώσω την, ε, τις προσδοκίες σας ε, και να ακολουθήσω και τα ίχνη της προκατόχου μου που κατά τη γνώμη μου έκανε εξαιρετική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Μοζέρα, Ντεπέ. Καλώς ορίσατε, κύριε Πίτροπε, και καλή επιτυχία. Γιατί ε, ξέρετε ότι έχουμε κάποιες ε, προτάσεις όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καινούργιο σύστημα. Αυτό που προτείνει το Κοινοβούλιο. Είπατε στην ε, απάντηση ότι η πραγματική πρόκληση είναι να φτάσουμε μια φάση κατά την οποία θα το δεχθούν τα κράτη-μέλη σε την του συστήματο. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει όμω καμία τέτοια περίπτωση εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαμορφώσει μια αξιολογή πρόταση. Και σα ερωτώ, ακόμα και αν αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, εσεί δεσμεύεστε όσον αφορά μια τέτοια πρόταση πριν την πρώτη η Πρώτου του 18 και αυτό είναι τα συστατικά ε, στοιχεία ενός καινούργιου ζητήματος ιδίων πόρων σύμφωνα με την ομάδα Μαντή. Επίσης ε, πρόσφατα η Κομισιόν καλέσει κάποια πρόταση για αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου και έτσι να υπάρχει μια κατανομή των προσφύγων στα κράτη-μέλη καινούριο τρόπο. Κάποια μέλη λένε ναι, κάποια λένε όχι και εσείς όμως ε, έπρεπε να ε, προβλέψετε κάποια πρόστιμα όσο δεν συμμορφώνονται και σας ρωτώ εσείς ε, αντί για πρόστιμα στο μέλλον δεν θα ήταν πιο λογικό να προβλέψετε να υπάρχει χρηματοδότηση των κρατών μελών από τα διευθυντικά ταμεία και έτσι να υπάρχει χρηματοδότηση των αναγκαίων μέτρων, ούτως ώστε να υπάρχει η καταγραφή, η ένταξη, η εκπαίδευση των προσφύγων. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Επίτροπε. Αξιότιμη κύριε Ντεπρέ, σας ευχαριστούμε για τις διαρωτήσεις. Ε, η την έκθεση Μόντι ε, χθε ε, τη διάβασα πρώτη φορά. Είναι εξαιρετική ποιότητα, ε, 90 σελίδε ε, και είναι κατάλληλη ε, χρονική στιγμή διότι χρειαζόμαστε μία εις βάθος διαπραγμάτευση για την κατάσταση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμάσουμε τα επόμενα δημοσιονομικά πλαίσια και χρειαζόμαστε νέα έσοδα. Και επίσης με το Brexit χρειαζόμαστε διαρθρωτικού τύπου αλλαγή στον προϋπολογισμό. Και η έκθεση και η Επιτροπή Μόντι είναι ε, κάτι που ε, δεν ζήτησε μόνο το Κοινοβουλίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προέκυψε ως ανάγκη από το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το, μέχρι το 2013 δηλαδή, και επισημάνθηκε αυτό από όλα τα θεσμικά όργανα. Ε, ε, δεν πάμε στην τύχη. Ε, ε, έχουμε επίγνωση του προβλήματος και θέλουμε να αναβαθμιστεί η διαδικασία. Υπάρχουν ε, προτάσεις για τον ενεργειακό φόρο, για το διοξίδιο του άνθρακα, ε, για το ΦΠΑ. Ε, αυτή η έκθεση θα είναι η βάση για μια ανοιχτή συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Για το Δουβλίνο Ξέρω πολύ καλά το πρόβλημα ε, των ποσοστώσεων και κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία για την υποδοχή προσφύγων, ε, για την οικοδόμηση κέντρων υποδοχής, ε, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών, κατά τη γνώμη μου. συγγνώμη που μακρηγόρησα. Κύριο κύριος Κέλμερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Έντιγκερ, που είστε εδώ στη θέση μα για ερωτήσει και απαντήσει. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για τον προπολογισμό. Ξέρουμε ότι του επόμενου μήνε θα αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Βρετανοί. Πολύ συγκεκριμένα, λοιπόν, θεωρείτε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και αν ναι, θα χρειαστεί να συμβάλλουν περισσότερο τα εναπομείναντα κράτη-μέλη ή θα πρέπει να περιοριστεί ο προπολογισμό. Και η δεύτερη ερώτηση, που είναι πιο γενική φύσεως, Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι και εσείς το πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπούμενη από τους επιτρόπους πρέπει εν όλο όργανο να φέρει και την ευθύνη για κάθε τι που είναι αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η θεσμοφύλακας των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές συχνές παραβιάσεις αυτών των συνθήκων. Συνθήκη του Μαστρίχτ, συνθήκη του Δουβλίνου, ε, από ό,τι φαίνεται δεν αξίζουν καν το χαρτί πάνω στο οποίο έχουν γραφτεί. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ένας κανονισμός καινούριο που αφορά τις τράπεζες που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην υπόθεση dei Paschi της Θελικής Τράπεζας. Και πάλι φαίνεται ότι θα υπάρξουν παραβιάσεις του σχετικού, των σχετικών διατάξεων. Κύριε Επίτροπε, εσείς συγκεκριμένα και προσωπικά τι κάνετε έτσι ώστε να ε, σταθείτε στο πιο των ευθυνών σας. Απάντηση οι κανόνες σχετικοί με την χρηματοπιστωτική κρίση, την οικονομική κρίση, όπως τους όρισε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, είναι ε, δεσμευτικοί για όλους. Αυτό αφορά το νέο χρέος, αφορά το συνολικό χρέος, αφορά τον τομέα των τραπεζικών, τον χρηματοπιστωτικό. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγουμε εντατικότατες ε, συνομιλίες και επαφές και ιδιαίτερα έναντι του Eurogroup και του Συμβουλίου εν όλο αλλά και του, και του Κοινοβουλίου με ε, αρμόδιο καθήλυνο τον συνάδελφο Ντομπρόφσκης αλλά και μεταξύ και των λοιπόν βεβαίω επιτρόπων, ιδιαίτερα στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η, Επιτροπή, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινείται πάντα μέσα στην ομιμότητα των ευρωπαϊκών συνθήκων με την ευελιξία που είναι δυνατή, μεν αλλά χωρί παραβίαση των ορίων. Και θα ήθελα να δώσω μια ακόμη πολύ σημαντική απάντηση για τη μελλοντική δημοσιονομική μας πολιτική, διότι ε, παρά την επιστροφή του, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει καθαρός χορηγό του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να κατατεθεί η πρόταση για την αποχώρηση από το Λονδίνο, ε, να προσδοριστεί το χρονοδιάγραμμα, να δούμε αν θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, τι είδους προτάσεις θα κατατεθούν. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα την απάντηση μπορώ να σα τη δώσω πολύ πιο ευχερός μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από ότι τώρα. Ε, θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα οποία δεν καλύπτει ω πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα τα καλύψουν τα άλλα κράτη-μέλη και πάντω θα αναστήσουμε τον πιο δίκαιο και μέσο δρόμο. Παρακαλώ, κύριε Στανά. Στη σημερινή συζήτηση δυστυχώς. Δεν έχουμε το χρόνο τόσο ώστε να γνωριστούμε καλύτερα. Αλλά ξέρω τον κύριο Άντζιπ, τον πρώην προϊσταμένο σα. Ε, ξέρουμε ότι έχετε πασχίσει για την ψηφική πολιτική και για τους ανθρωπινούς πόρους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής με τον προπολογισμό. Πρόσφατα το ελληνικό συνέδριο είπε ότι έχουμε αποτύχει να καλύψουν τον προπολογισμό την αλλαγή του κλίματος. Άρα, σας ερωτώ εσείς τι πιστεύετε και τι θα προτείνετε εν ώψη της χρήσης του 2018 και όσον αφορά την του του δημοσίου πλαισίου σε σχέση με αυτό το θέμα, την αλλαγή του κλίματος. Θα σας απαντήσω κύριε Βρεφτά ότι η συνεργασία μου με τον κύριο Άντζιπ ήταν εξαιρετική και σε φιλικούς όρους καταρχάς. Δεύτερον, είχα την ευθύνη δύο γενικών διευθύνσεων. Προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλα ζητήματα δικαίου ή ζητήματα της εσωτερικής αγοράς ή ζητήματα του ανταγωνισμού ήταν θέματα τα οποία ε, προχωρούσαν σε συντονισμό υπό τον Αντιπρόεδρο και κοινή συνεργασία και ευθύνη. Για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές το Κοινοβούλιο νομίζω ότι έχει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για την επιτυχία της διασκέψεως των Παρισίων με αποτελέσματα τα οποία τουλάχιστον είναι εφικτά. Στον ευρωπαϊκό προπολογισμό έχουμε ένα στόχο του 20%. 20% των επενδύσεων και των δαπανών που θα πρέπει να είναι αφιερωμένες στο ε, θέμα της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να το ποσοστικοποιήσουμε αυτό συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται για μια πολιτική δέσμευση και μια στόχευση. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως το 20% είτε πρόκειται για ε, υποδομές, για προγράμματα συνοχής, για ε, γεωργία, για πρασίνισμα, για εκτακτικοποίηση στην παραγωγή, είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και στι τωρινέ μου αρμοδιότητε, ε, το θέμα των κτηρίων είναι παραδείγματι του Λουξεμβούργου και των Βρυξελών, που ήδη έχουν, ε, έχει απασχολήσει του προκατόχου μου. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση, ώστε να εξασφαλίσουμε και από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετοχή στον περιορισμό των ε, ενεργειακών δαπανών ευχαρισμό από την ομάδα ΕΝΕΦ έχουμε έναν ομιλητή που όμως δεν μας έχει δώσει το όνομα συγκεκριμένα του βουλευτή που θα λάβει το λόγο. Ποιος βουλευτής σκοπεύει να λάβει το λόγο εκ μέρους της ομάδας ΕΝΕΦ. Δεν βλέπω εκπρόσωπο. Η κυρία Νίριαντα λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βεβαίω και ο Επίτροπο Χρυσέ με τις, ε, το θέμα των ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Όμω είναι πάρα πολύ εύστοχο το πολιτικό κλίμα. Οπότε με αυτή την πολιτική αστάθεια που η κυριαρχή και όλε αυτέ τι κρίσει μα έχουν χτυπήσει και ότι συνέχεια υπάρχει δυσάρσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ βλέπετε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτή την τρική μία. Μιλήσατε για ισότητα, αλλά επίση μα είπατε ότι έχετε πει ότι ε, μετά τα 40, ε, στα 40 έχει φτάσει κάποιο στην μέγιστη απόδοση και μετά οι μεγαλύτεροι δεν αποδίδουν κλπ. Μα, τι, θα, τι, τι, λέτε για αυτά. Πρέπει να μας διαβεβαιώσετε σχετικά, γιατί πώς θα μπορέσετε έτσι να επιβάλλετε διαφάνεια και ηθική, πώς πώς μπορείτε να μας ε, ε καθισχάσετε ότι όλα αυτά τα φέρετε εις πέρας και με τον σωστό τρόπο. είναι ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα με έχει ήδη απασχολήσει. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τις εργασίες ε, της ε, γενική Διεύθυνσης για την Ενέργεια, της Κολέκτερα και άλλες. Μπορείτε απλώ να ρωτήσετε, μπορώ να σα απαντήσω βεβαίω, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και τι πολλέ χιλιάδε εργαζομένου και τι βάδε Βιτεμβέργη, όπου είχα τι ευθύνε κι εγώ ω υπάλληλο. Επίσης, εκεί μπορέσαμε να περιορίσουμε για τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους το χρόνο εργασίας, εβδομαδιαίες εργασίας, κυρίως για τους ε, διδάσκοντες, για τους δασκάλους άνδρες και γυναίκες, έτσι ώστε να περιορίσουμε και την ε, επιβάρυνση σωματική, ε, επιβάρυνση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα burnout. Θα μπορούσε ένα δάσκαλο βεβαίω να εργάζεται μέχρι το, τα 55 του και τα 65 του με λιγότερε όμω ευθύνε. Αυτή ήταν η προσέγγιση μας η οποία οδήγησε σε περιορισμό τη εβδομαδιαίας απασχόλησης και αντίστοιχα μικρό περιορισμό του μισθού που ήταν προς το συμφέρον και των ίδιων των εργαζομένων για διαφύλαξη της ε, σωματικής τους υγείας πάνω απ' όλα και της αποδοτικότητάς τους. Η ευθυντή έχει τρία λεπτά για να θέσει την ερώτησή του. Αλλά ούτε εσεί μα εγνωρίσατε το ποιο θα λάβει το λόγο. Υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο ομάδα που θέλει να ε, υποβάλει την ερώτηση. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Οπότε το λόγο έχει ο κύριο Άλμπερ. Κύριε Επίτροπε, η Επίτροπος Γεωργίευα συνήθως υποστήριζε τις θέσεις μας και έρχονταν εδώ να τα πούμε. Δεν θεωρώ ότι εσείς θα έρχεστε ακόμα συγχρονότερα. Τώρα έχω στις υποβάλει τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το πολιτές πλαίσιο. Ξέρουμε πώς έγινε η αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου ε, και θα ακολουθήσει τώρα η αναθεώρηση του μέλος πλαισίου. Οπότε για πέστε μου, άπαξ και αρχίσουμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά το επόμενο για σημείο Πότε θα γίνει αυτό και πότε θα ολοκληρωθούν πάνω κάτω. Πέστε μας τι, τι timing θα διευθεί η διαδικασία. Άλλη ερώτηση όσον αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Ε, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τους αιτήσους προπολογισμούς. Άρα εσείς πώς το Κοινοβούλιο όσον αφορά την προπαρασκευή αυτού του ε, πολιτού ε, πλαισίου. Να μην έχουμε κάποια διαδικασία κοινή ad αλλά να γίνει μια άρτια προπαρασκευή. Επίτροπος. Το κοινοβούλιο είναι ένα, ένας συνομοθέτης απόλυτα σεβαστός με πλήρης αρμοδιότητες μαζί με το Συμβούλιο. Έχουμε ένα ένα νοσονομικό πλαίσιο που εκπνέει το 2020, το 2020. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις να πούμε ότι εάν το Brexit αρχίσει να ισχύει από το 2019, θα έπρεπε να περικοπεί η διάρκεια του πολιτού δημοσιονομικού σχεδίου. Ωστόσο, εγώ είμαι επιφυλακτικό στην αντίμεση τη πρόταση. Οι ειδικοί με του οποίου έχω συνομιλήσει από το επιτελείο μου λένε ότι αυτό εμπεριέχει σημαντικού κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, μέχρι το τέλο του 2017 θα ετοιμάσει τι δικέ τη προτάσει για το προσεχέ πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα πρέπει να συνομιλήσουμε λοιπόν ε, με τους Βρετανούς, μαζί σας μάλλον για να δούμε αν θα είναι επταετές, αν θα είναι πενταετές και να εμβαθύνουμε στα ζητήματα. Ε, πότε ακριβώς θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ε, θα απαντήσω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν είναι και πιο ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα για το Brexit, για να δούμε ακριβώς πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές για το προσεχές πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να κοιτάξουμε και την νεολαία μας. Η προσεχής επιτροπή επίσης θα είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να έχει την τελική ε, λέξη, όπως άλλωστε και το προσεχές κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2019 και το Συμβούλιο αντίστοιχα. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ε, παράδοση, παραλαβή της σκητάλης στην περίοδο αυτή του 2019-20. Δεν μπορώ να προκαταβάλω λοιπόν ε, θέσεις και ιδέες, είτε σε επιτροπές, είτε σε συνομιλίες. Όποιος με γνωρίζει από την Επιτροπή ΙΤΡΕ τα τελευταία, 7 χρόνια ήμουν πάντοτε διαθέσιμος για να δίνω απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών. Πολλές φορές μάλιστα προκαταλάμβανα ε, προβληματισμούς δικούς σας και ζητούσα εγώ να έρθω να μιλήσουμε σε θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ κύριο Βιώτη, έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ήδη συζητήσαμε για τους ανθρώπινους πόρους και συζητήθηκαν και οι δηλώσεις οι οποίες ε, προέβεται όσον αφορά τους ε, ΛΟΑΔ. Οπότε θα πρέπει να πούμε όμως περισσότερα γιατί έχουμε αυτή την απάντησή σας που μιλάει για αυτή τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη όσον αφορά το σημείο για τους ΛΟΑΔ. Μήπως θα μπορούσατε να μας τα πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα ακριβώς εσείς τι προτάσεις θα κάνετε όσον αφορά αυτό. Τι γίνεται επίσης με τα ζεύγη ε, των ε, προσώπων ιδίου φίλου, τι γίνεται επίσης με τους δύο εμφυλικούς. Έχουμε τις σχετικές ε, δηλώσεις αλλά πες μας τι θα ακολουθήσει. Κύριε Βουλευτά, γνωρίζω ότι η Επίτροπος Γεωργίευα είχε με τους δικούς της ε, συναδέλφους και με βουλευτές πολλές φορές συνομιλήσει ε, στα θέματα που σας απασχολούν και είχε προσδιορίσει άξονες εργασίας που ολοκληρώνονται στους επόμενους μήνες για να προσδορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα που θα εξασφαλίσει και καλή ποιότητα προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα μόνο. Θα πρόκειται λοιπόν για την ε, εφαρμογή της περικοπής του προσωπικού κατά 5% που πρέπει μέχρι το 2017 να υλοποιηθεί. Ε, εδώ θα έχουμε να κάνουμε και με την ανάπτυξη προσωπικού στελεχών μέσων ή ανώτερων ε, γυναικών και αυτό σταδιακά θα σημάνει την υλοποίηση των στόχων έως το 2019. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα αποτροπής των διακρίσεων σε επίπεδο όλης της Επιτροπής εναντί ουδήποτε και ιασδήποτε υπαλλήλου. Σε αυτό θα συμβάλλουμε. Έχουμε να κάνουμε επίσης, γιατί αναφέρθηκε και η Όλαφ, με, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τις εκθέσεις που είναι γνωστές της πάση. Και ήδη έχει η κυρία Γεωργίευα αναλάβει αυτό το έργο και θα το συνεχίσω εγώ. Ευχαριστούμε λίγο. Πρώτα τώρα η δική μου πολιτική ομάδα. να σας προβάλλω την ερώτηση. Ότι είχατε αναλάβει τον προϋπολογισμό. Είπαμε ότι μιλά στον πολίτη αυτός ο ολός και με το κείμενο το οποίο όμως τελικά δεν λέει τίποτα στον πολίτη. Υπήρχε ένα πλαίσιο πάρα πολύ στενό, μιλούσαμε για πολιετή χαρακτήρα, μιλούσαμε για, για κονδύλια και μέσα στην κρίση είπαμε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν καινούργια μέσα πολιτικής. οπότε μιλήσαμε για την καρδιά του προπολισμού, για έναν γαλαξία δημοσιονομικό αλλά υπάρχουν και οι σχετικοί δορυφόροι που είναι πολύ και με την Γεωργίευα συζητήσαμε για το πώς είναι δυνατόν μπορεί να είναι κατανοητός ο προϋπολογισμός στον κόσμο. αν θέλουμε να έρθει κοντά στον κόσμο η Ευρώπη θα πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος στην Ευρώπη αλλά και τον προϋπολογισμό. Εσείς πώς θεωρείτε ότι αυτό θα υλοποιηθεί, πώς θα καταφέρουμε η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε κάποιον κατανοητό από τον κόσμο προϋπολογισμό. Πρόεδρε, μου δώσατε την γραφική παράσταση αυτή με το γαλαξία, το μελέτησα και μιλήσατε για αυτούς τους δορυφόρους ε, ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι στο κέντρο, αλλά υπάρχουν ε, καταπιστεύματα, διάφορα νέα μέσα, ε, νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ε, διακυβερνητικά ταμεία που τελικά περιορίζουν τρόπον την, τις δυνατότητες που δικαιωματικά κατέχει το Κοινοβούλιο. Αυτή η συζήτηση θα γίνει στα πλαίσια τη αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Πάντοτε ε, έρχονται στιγμές που χρειαζόμαστε εξωτερικά εργαλεία. Όμως, ε, μεσοπρόθεσμα, ε, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εσωτερικοποιηθούν τα νέα μέσα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στα όρια αυτού του νέου γαλαξιά και ε, ναι, προτίθεμε να συζητήσουμε για αυτά τα νέα μέσα, αλλά μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να ενταχθούν στον προπολογισμό, ούτω ώστε να μπορέσετε κι εσεί να υπομειστείτε τι πολιτικέ ευθύνε και να ενισχύσετε το δημοκρατικό σα έλεγχο. Ε, θα μιλήσω ειλικρινά. Ε, Νομίζω ότι δεν επαρκούν αυτά που κάνουμε να τα λέμε μεταξύ μας. Κάθε δήμαρχος, κάθε υπάλληλος της δημόσιας διοίκησης, ο καθένα θα πρέπει να διαπιστώσει ποια είναι τα ωφέλη του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά που συμβαίνουν σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Τα συνδικάτα, ε, οι εργαζόμενοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν διότι ε, είναι πολύ σημαντική η εισφορά του προπολογισμού για τη λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς για την καταπολέμηση τη διαφθοράς ενέσχυση της ανταγωνιστικότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερου εταιρού σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι συμφωνείτε με το θεματολόγιο της κ. Γεωργέβα όσον αφορά έναν προπολογισμό που να στοχεύει σε αποτελέσματα. Για πέστε μας, ε, επικτηνόμενος πάνω σε αυτό, πώς θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει το πολιτές δημοσιοκοπλαίσιο και τη σχετική προβληματική. Δεύτερον, η κυρία Γεωργιέβα εξήγηλε μία ανώτερη θέση υπαλλήλου που θα είναι αρμόδιος να ελέγχει την απόδοση, τις επιδόσεις των σπάντων του προϋπολογισμού. Πώς ποτέ να καλύψετε αυτή τη θέση και πότε. Ε, φυσικά προτίθεμαι να ε, φροντίσω ώστε να πληρωθεί αυτή η νέα θέση ε, Τώρα, αυτή η ιδέα να προσανατολιζόμαστε στα αποτελέσματα, δηλαδή να εστιάζεται ο προπολογισμό στα αποτελέσματα και σε επιδόσεις, είναι μια ιδέα που βρίσκω λογική και θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι επενδύσεις μας, ε, να προσμετρούμε την αποτελεσματικότητα των δαπανών μας. Η έκθεση Μόντι μιλάει για την προστιθέμενη αξία ε, και σε αυτό μένει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πώς αποτελεσματικότερα, με λιγότερες δαπάνε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μπορούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις. Ε, ευσταθεί η επιχειρηματολογία μας είναι περιστατωμένα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε και άρχισα να κάνω ε, τις επαφές με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Θα συνεχίσω ε, στο Λουξεμβούργο, ε, διότι παραμένει ψηλό το ποσοστό των λαθών ε, προς πρόσθετες πράξεις ε, θα πρέπει να θεσπίσουμε, όχι εναλλακτικέ. Νομίζω ότι η ενίσχυση των ελέγχων, ε, ε, ταυτόχρονα με την ενίσχυση των αξιολογήσεων, είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Και επίσης η εμπειρία σας είναι πολύτιμη από την εκλογική σας περιφέρεια. Ξέρετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ποια είναι, ποια είναι η αποτελεσματικότητα, ποια είναι τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Και αυτή την εμπειρία σας θέλουμε να την εξοπλίσουμε και εμεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εστεμπάν Γκονσάλες Πόνς. Ευχαριστούμε κύριε Ότιγκερ και πρώτα πρώτα συγχαρητήρια για το βιογραφικό σας που ακριβώς δείχνει ότι ο κατάλληλο πρόσφυγε για κατάλληλη θέση αλλά εδώ υπάρχει κάτι το οποίο έχει σχέση με το κατά πόσο εμείς τηρούμε τις αρχές μας. Πρόκειται για το προσφυγικό ε, που έχει δημισιονομικές συνέπειες. Είναι γεγονό ότι έχουμε πάρα πολλέ υπηρεσίε και έπρεπε να αλλάξουν την πολιτική του, ή ε, την πορεία του ε, πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια. Άρα, ε, πώ το βλέπετε σε πλευράς νομική το προσφυγικό και την πολιτική που ασκεί από αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, με ποιο τρόπο εσεί θεωρείτε ότι θα πρέπει να πολιτευτούμε από αυτού άμεσα επόμενα χρόνια. Επίσης, πώς θα έρθει αυτή η αντίφαση του ότι να έχουμε όλο ένα και περισσότερες ανάγκες όσον αφορά το προσφυγικό και από την άλλη όμως να έχουμε λιγότερες ζωέ. Για τους πρόσφυγες τα ε, κάποια κράτη-μέλη, η Ισπανία ε, παραδείγματος χάρη από το 2009, ε, η Ιταλία για τη Λαμπεντούσα ήδη πριν από πέντε χρόνια είχε αναγνωρίσει το πόσα έπρεπε να γίνουν για τους πρόσφυγες. Λοιπόν, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, ακόμη και τα κράτη-μέλη που δεν βρίσκονται στη Μεσόγειο θα πρέπει να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορώ να μιλήσω για τη χώρα μου. Ε, μια, η μεγαλύτερη χώρα. Άργησε να αναγνωρίζει τη σημασία της αλληλεγγύης ε, ως προς την προσφυγική χρήση. Ε, τα τρία θεσμικά όργανα άρχισαν μόλις πρόσφατες σοβαρέ διαπραγματεύσεις και αυτές θα πρέπει να τις συνεχίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος από κοινού να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ο Frontex είναι πολύ μικρός οργανισμός, δεν επαρκεί. Ε, το Σέγγεν, το Δουβλίνο ε, δεν επαρκούν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέους ε, ανθρώπινους και οικονομικούς οπόρους ώστε να ενισχύσουμε τη δράση προστασίας των συνόρων, προστασίας των ατόμων. Ε, για την υποδοχή των ε, προσφύγων, για την επεξεργασία των αιτήσεων. Η, η Ελλάδα ε, για την διοίκηση, για την διαχείριση των αιτήσεων δεν μπορεί να από μόνη της να αναλάβει αυτό το έργο. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την Ιταλία, για την Βουλγαρία. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι για την προσφυγική κρίση θα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα κράτη-μέλη. Ε, ε, από την Ιγυρία, από το Μάλι, από την Αίγυπτο έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν προοπτικές στη χώρα τους για παραμείνουν εκεί πέρα. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τις υποδομές σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο κοινοβούλιο εμείς. Ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το έργο του και το μελλοντικό κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Γιάννη Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη σημερινή ακρόαση αναφέρθηκε ήδη αρκετές φορές η επικείμενη αναθεώρηση του του δημοσιονομικού πλαισίου και έχουμε επισημάνει κάποια ζητήματα. Ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν αντίστοιχα το ρόλο τους στις ε, διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ποια είναι η κατάσταση. Διαπραγματεύονται τελικά τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και δεν μιλάμε για το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, ε, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, προσπαθούν να βρουν την καλύτερη οικονομική λύση για αυτού, δηλαδή πώ μπορούν να περιορίσουν στο ελάχιστο τι εισφορέ στον προπολογισμό για τη διαχείριση αυτού του προβλήματο. Ε, αναμεταδίδεται η συζήτηση, θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ώστε να μην χειροτερεύσει η κατάσταση για τους φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έτοιμη η έκθεση μόντε. Δυστυχώ ε, δεν ε, είχα τη χαρά να τη διαβάσω. Ε, Χάρηκα με αυτά που είπατε, φυσικά θα τη διαβάσω, αλλά θέλω στο μεταξύ να μου πείτε, κατάλαβα καλά, ε, θέλετε ε, μέσω μακροπρόθεσμα για το ε, πολιετές ε, δημοσιονομικό ε, πλαίσιο τελικά να συνδυάσετε ε, τις διαπραγματεύσεις με πρόταση για νέους ιδίους πόρους, αυτό είπατε. Ναι, μπορώ να απαντήσω σύντομα. Ναι, αυτό είπα. Ε, ιδανικά θα πρέπει ε, φέτος να ετοιμάσει την πρότασή της για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μότιος, πρώην Πρωθυπουργός, ε, έχει κύρος στο Συμβούλιο και ε, σε στο Κοινοβούλιο το ίδιο, αλλά έχει και τι επαφέ του στην Επιτροπή. Είναι λοιπόν μια κατάλληλη χρονική στιγμή την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ο στόχος δεν είναι να αυξηθεί η εισφορά των φορολογουμένων. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσουμε τα θεμέλια αυτού του προϋπολογισμού που ε, λειτουργούν μονομερώς για κάποιους τομείς μέχρι στιγμής. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όλοι οι επίτροποι στη χώρα τους ε, θα πρέπει να στον τομέα της αρμοδιότητάς του να αγωνιστούν και εμείς το ίδιο. Ε, εγώ ελπίζω ε, να μας βοηθήσει ο Μάρτιν Σούλτ ως μελλοντικό μέλος της ε, γερμανικής κυβέρνησης. Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Σόιμπλε, με την κυρία Μέρκελ. Εάν ε, η χώρα μου με βοηθήσει, αν το ίδιο ε, κάνουν και άλλες χώρες για τους ε, επιτρόπους τους, ε, δεν θα παραμείνει στο σιρτάρι η έκθεση Μόντι και θα χρησιμεύσει σε κάτι. Ευχαριστούμε κύριο Πόλη Ρουμπίκ τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια κύριε Έτεγκερ για τη δουλειά που έχετε μέχρι τώρα επιτελέσει. Σας γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια στην Επιτροπή βιομηχανία, ήσταν πάντοτε στη διάθεσή μας με πολύ αρμόδια, κατάλληλη και σωστή ενημέρωση. Η δουλειά του Επιτρόπου σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει αποτελεσματικότητα και εμείς βεβαίως ως Κοινοβούλιο ιδιαίτερη αξία που δίδουμε και το έχουμε δείξει και στις διάφορες συνομιλίες μας ε, στην ε, συνδιαλλαγή τον ορίζοντα 2020, την, ε, το θεματολόγιο για την έρευνα. Έχουμε λοιπόν προσδορίσει τις προτεραιότητές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν τώρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το σχετικό πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την ε, έμφαση που θα πρέπει να δοθεί και την ενίσχυση του προγράμματος, όπως επίσης και το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες, που είναι από τα πιο επιτυχημένα μας προγράμματα. Πρέπει να διεθνοποιηθεί τώρα πια, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε και νέα πρότυπα για τους νέους επιχειρηματίες που θα δημιουργήσουν και στην Ευρώπη αλλά και με τη διεθνή τους εμπειρία νέες θέσεις εργασίας. Ποιες ευκαιρίες λοιπόν διαβλέπετε εδώ για το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο γιατί ξεκινούν τώρα οι διαπραγματεύσεις με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ποια είναι η δική σας ε, έποψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ε, δραστηριοποίησή τους στο διεθνή πλέον, ε, στο διεθνές σκηνικό. Απάντηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό έχουμε δύο κεφάλαια ιδίω, τα οποία ορίζουν το, τη βάση της χρηματοδότησης και της υποστήριξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα α ιδιαίτερος είναι το κεφάλαιο το οποίο ε, δίνει έμφαση στην καινοτομία με το Erasmus Plus για την ε, νέα γενιά, με τα προγράμματα για την απασχόληση των νέων εν γέννη με τα προγράμματα υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των ε, ε, startups, ε, των νεοφυών επιχειρήσεων και αντίστοιχα άλλα προγράμματα. Στον τομέα τη ψηφιακή οικονομία τα τελευταία χρόνια μπορούσα να συλλέξω πολύτιμη εμπειρία, ιδιαίτερα για την ε, προστιθέμενη αξία, για την πολύτιμη προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η ευρωπαϊκή διάσταση, ιδιαίτερα στη μικροτεχνολογία και την ανοτεχνολογία, του σένσορε, τα, τη ρομποτική. Έχουμε πολύ σημαντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Έχουμε ε, συνεργασίες, joint undertakings και κυρίως έχουμε να κάνουμε με την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία μεταξύ διαφορών κρατών. Κανείς μόνος δεν μπορεί να τα καταφέρει όλοι μαζί, όμως μαζί και με το βιομηχανικό κλάδο και με τους ερευνητές μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Και σε σχέση με τις ΗΠΑ, τους ανταγωνιστές μας και με τους ανταγωνιστές βεβαίως της Ασίας. Ε, ξέρετε βεβαίως ε, ότι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, η Νότια Γερμανία, δεν έχει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ένας τομέας που γνωρίζω πολύ καλά και έχω ε, δεσμευθεί να υποστηρίξω. Ευχαριστώ, κύριος Μας, Μάνκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η απασχόληση των νέων συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό 2016 στη διαδικασία της συνδιαλλαγής δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσουμε νέα κονδύλια για την απασχόληση των νέων. Και έτσι ήταν ε, ήδη γνωστό πως υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Είχαμε κάνει τότε μία δήλωση όπου ιδιαίτερα καλούσαμε τα κράτη-μέλη έως το 2015 να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του προγράμματος για να ληφθούν στη συνέχεια οι αποφάσεις. Η αξιολόγηση ωστόσο κράτησε 10 μήνες αντί για 3 εβδομάδες. Αν και θα είχαν αρκέσει οι 3 εβδομάδες. Χάθηκε ένας χρόνος ολόκληρος λοιπόν για την αξιολόγηση αυτήν από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους ε, καταγράφεται μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία του προγράμματος με ένα τρίτο ε, της ανεργίας των νέων, ε, με μείωση δηλαδή κατά ένα τρίτο της ανεργίας των νέων, 500 εκατομμύρια που μπόρεσαν να ε, υλοποιηθούν ως κονδύλια και τι είχε ζητήσει περισσότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. Κύριε Επίτροπε, τι σκοπεύετε να κάνετε για την απασχόληση των νέων για το έτος 2018 και την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου έτσι ώστε η σημαντική αυτή προτεραιότητα να μην λησμονηθεί και πάλι. Απάντηση. για την ε, αναθεώρηση του πολιτισμού συνομικού πλαισίου. Πρέπει πλέον να δώσει το πράσινο φως στο Συμβούλιο ώστε να ξεκινήσουν οι ε, συνομιλίες ε, με συγκεκριμένα στόχους μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Μαζί με όλους τους συναδέλφους λοιπόν της Επιτροπής έχουμε πολύ συγκεκριμένα και καλά επιχειρήματα προβάλλει στο Συμβούλιο και εξηγούμε ότι η απασχόληση των νέων και τα σχετικά μέτρα είναι αποτελεσματικά έχουν ήδη καταγράψει τα πρώτα θετικά βήματα στην αγορά εργασίας και πρέπει να συνεχιστούν. Είμαι βέβαιος μάλιστα ότι η αγορά εργασίας, οι αγορές εργασίας στις διάφορες περιοχές ε, της Ευρώπης μπορούν χάρη στο Youth Employment να έχουν πολύ ε, θετικά αποτελέσματα στην επόμενη περίοδο και μετά δηλαδή το 2020. Και βεβαίως μπορούμε να επιτύχουμε μόνο αυτό που δημοκρατικά είναι εφικτό. Ε, αυτό δηλαδή που μπορώ να δεσμευθώ είναι ότι κάθε ευρώ που θα έχουμε στη θέση μας θα αξιοποιηθεί κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και βεβαίως ότι σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα αγωνιστώ όσο περισσότερο μπορώ στις συνομιλίες με το Συμβούλιο για καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Σέλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε κύριε ε, την για την ε, εισαγωγή σας ομιλία. Κύριε Επίτροπε, στην σημερινή συγκυρία έχουμε λαϊκισμό ε, στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι έχουμε ε, κάποιους πολιτικοί πολιτική η οποία ε, είναι και περίεργη. Είναι σουρεαλιστική, οπότε θα πρέπει να δούμε τι είδους προγράμματα θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση όσον τον πολιτισμό, γιατί αυτό, αυτό είναι η λύση. Είναι το κλειδί ούτως ώστε να εξηγηθεί στον κόσμο τι πάει να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να έρθει πιο κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Να έχουμε κάποια προγράμματα ούτως ώστε και συναισθηματικά να δεθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ευρωπαίοι. Α πούμε το Europe for Citizens είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εσεί, πώς το βλέπετε και πώς επίσης θα άρετε αυτή την αντίβαση μεταξύ του ότι θέλουμε να υπάρχει περισσότερη χρηματοδότηση για τα σχετικά προγράμματα και από την άλλη μεριά ε, την ε, πραγματικότητα. Γιατί έχουμε το τρίτο κεφάλαιο που λέει για την ιδιότητα του πολίτη, λέει για την ε, ασφάλεια και εκεί δεν έχουμε από αποθεματικό. Ευχαριστώ για την απάντησή σα. Επίτροπο. Ένα τμήμα των προγραμμάτων που εσείς ε, αναφέρατε ήταν στις αρμοδιότητές μου τα προηγούμενα χρόνια. Ε, νέα μέσα, ε, πολιτισμός και άλλα διάφορα, όπως όμως είχε και ο συνάδελφος Νάφρατσιτς αντίστοιχα θέματα στην αρμοδιότητά του. Νομίζω λοιπόν ότι τα διαστροτικά, η συνοχή, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η γεωργία, οι υποδομές, η έρευνα έχουν ένα μεγάλο κορβανά ούτως επί από τον οποίο όμως μπορούμε να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά έργα. Εάν έχουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως εκ τούτου, με σχετικά περιορισμένες δαπάνες, με λίγους πόρους, μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και κατανόηση για την Ευρώπη σαν αποτέλεσμα. Αυτό σε συνεργασία λοιπόν με το Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με εσά, μπορούμε να το, να το αναπτύξουμε, να οικοδομήσουμε πάνω στην εμπειρία δηλαδή που έχουμε και να προχωρήσουμε σε πιο καλά αποτελέσματα, χωρίς να μιλούμε για δισεκατομμύρια απαραίτητα. Με ένα εκατομμύριο με λίγα χρήματα μπορούμε να έχουμε πολύ αποτελεσματικά προγράμματα για τον πολιτισμό, για την νεολαία, για την απασχόληση. Ευχαριστούμε λίγο, Πρόεδρος. Τον ε, λόγο έχει η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις τομείς πολιτικής όπου έχει δεσμευτεί να τους εντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προπολογισμό αλλαγή κλίμακος, βιοποικιλότητα και ισότητα των φύλων. Και αυτή η τελευταία πολιτική έχει προχωρήσει λιγότερο. Έχουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία για τι άλλε πολιτικέ, οπότε είναι δυνατόν το mainstream να γίνει σε σχέση με τον προπολογισμό. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν γιατί επένδυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να προχωρήσει αυτέ τι πολιτικέ. Όμω ε, το θέμα είναι τι γίνεται για τη μενισότητα των φίλων. έχετε αφιερώσει χρόνο αλλά και ανθρώπινου πόρου. Εκεί δεν προχωρήσαμε. Είσαστε υπέρ του να ενταχθούν στον προπολογισμό ε, αυτές οι πολιτικές, κυρίως η ισότητα των φύλων, και να έχετε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία όσον αφορά την κάλυψη από τον προπολογισμό της πολιτικής ισότητας των φύλων. Επίτροπος. Βεβαίως, πολιτικά είναι σημαντικό τα σχετικά κεφάλαια ενός προϋπολογισμού και τα επιμέρους προγράμματα να καλύπτονται. Και πέραν των διευθυντικών ταμείων, των ερευνητικών προγραμμάτων, του greening της γεωργίας, της υπαίθρου, να έχουμε οριζόντιους κοινού στόχους. Με το 20% των δαπανών, παραδείγματι, για την ε, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αλλά δεν είναι απλό αυτό. Στην ενσωμάτωση της του φύλου, gender mainstreaming, έχουμε πάνω απ' όλα να, κάνουμε, να, να δώσουμε και το καλό παράδειγμα. Εάν δούμε τη δομή του ε, προσωπικού, του οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους είναι γυναίκες. Σε καθήκοντα, γραμματέως, ε, βοηθού και κατώτερα γενικά ε, ανώτερε θέσει έχουμε συντριπτική πλειοψηφία γυναικών. Στα μέσα και ανώτερα στρώματα έχουμε ένα ποσοστό περί το 30% σε γυναίκε. Ο στόχο λοιπόν του 40% είναι ένα καθοριστικό στόχο για την Επιτροπή Juncker. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωση και γενικά ο τρόπος διατύπωση των συμβάσεων κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει τη διάσταση του φύλου. Εμεί θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι γυναίκες είναι μεγαλύτερο κομμάτι με την έννοια ότι έχουν 3-4 ε, χρόνια περισσότερα εργάσιμα χρόνια από ότι οι άντρες συνάδελφοί τους. Τα δημογραφικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία καλύπτουν αυτή τη διαφορά. Και έτσι, χωρίς να έχω καταλήξει σε μια συγκεκριμένη ε, απάντηση, μελετώ γενικότερους στόχους για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που θα σημάνουν την ενσωμάτωση του φίλου, την εξορρόπηση της εκπροσώπηση των φύλων και εμείς βεβαίω βεβαίως ε, αν έχετε κάποιες προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε. Ευχαριστώ. Κύριο Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Ο Γιένς Γκάιερ και ο Ζεράρντε έχουν ήδη θέσει τη δική μου ερώτηση, αλλά θα την διατυπώσω κάπως διαφορετικά. Θυμάμαι από την εποχή που ήμασταν μαζί στην Επιτροπή ότι είχατε μια αρκετά ρεαλιστική και πραγματιστική στάση. Καθαρά πρακτικά λοιπόν. Βλέπεις ότι τα ίδια, οι ίδιοι είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταρρυθμίσουμε πραγματικά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Γιατί πρέπει να πω ότι η θεώρησή μου δεν ήταν τόσο αισιόδοξη. Ίσως η περίοδος αυτή του Brexit να αποτελέσει και μια μεγάλη ευκαιρία. Θα ήθελα όμως μια ρεαλιστική απάντηση και όχι μόνο ευχολόγιο. Παρακαλώ. Απάντηση. Η έκθεση Μόντι δεν δίνει αυτοματισμούς για την εξασφάλιση περισσότερων πόρων. Οι περισσότεροι πόροι, ενίσχυση των πόρων συνεπάγονται και περισ... Ε, ενίσχυση της αιτιολόγησης. Πρέπει να καλυφθούν με τα σχετική αιτιολόγηση και βεβαίως ισοδυναμούν και περισσότερες επενδύσεις επί Ευρώπης. Μια σκέψη μόνο θα αναφέρω η μετανάστευση, η προστασία των συνόρων, η αναπτυξιακή βοήθεια για να αποτρέψουμε μεταναστευτικέ ροέ στο μέλλον πρέπει να γίνει ή αν γίνει τέλο πάντων καθήκον ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να επιβαρύνει ή να τραβήξει χρήματα από τον προπολογισμό της έρευνας ή από κάποιο άλλο τομέα. Εάν θέλουν τα κράτη να προστατεύσουν την Ευρώπη, έχουμε προφανώς επιχείρημα για να ζητήσουμε πεστρούς πόρους, χωρίς να πληγεί η ύπεθρος, η ανάπτυξη, η έρευνα, υποδομές ή οτιδήποτε άλλο. Ένα επιχείρημα λοιπόν σοβαρό για ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού συγκεκριμένη που θα είναι προς όφελος και των κρατών μελών των ίδιων και της ασφαλείας τους. Δεύτερον, η έκθεση Μόντι καταγράφει όλες τις δυνατότητες για ίδιους πόρους, με το σύστημα των ανταλλαγών ε, εκπομπών, το ETS, με φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, φόρο στο διοξίδιο του άνθρακα, φορολογία της ενέργειας, ε, σταθεροποίηση και διευκρίνηση των ποσοστών ε, του συντελεστή φόρου προσθεμένης αξίας. Όλα αυτά τα καταγράφει ως δυνατότητες και δεν μπορούν βέβαια να απορριφθούν ε, ανεφετέρου όλε αυτέ οι προτάσει. Ρεαλιστική λοιπόν πρόταση θα ήταν κάποιε από αυτέ τι προτάσει να γίνουν δεκτέ από το Συμβούλιο και έτσι να προχωρήσει η υπόθεση εδώ ε, δημοσιονομικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Νεκρέσκου. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε, Επίτροπε. Στην Ανατολική Ευρώπη Θέλω, θέλαμε να μάθουμε από εσά το εξή. Πρόκειται για την πολιτική συνοχή. Πώς βλέπετε το θέμα στα πλαίσια του πολιτού δημοσίου πλαισίου αλλά και του επομένου πλαισίου και τι θα γίνει με τους ε, πόρους που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί. Πώς το βλέπετε, πώς είναι εδώ να βοηθηθούν τα κρατημέλη τα οποία δυσκολεύονται σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Τώρα και κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Μιλώ για τις δηλώσεις του 2013 και σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας σας ότι αντί να καταπολεμήσετε την ε, κρίση προσπαθείτε ως χώρα να κουνήσετε το δάχτυλο, να, να εκπαιδεύσετε τον υπόλοιπο. Και μιλώ για Βουλγαρία, Ρουμανία και Ιταλία. Είπατε ότι η Γαλλία δεν είναι οικονομικά έτοιμη για να κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει όντως θεωρείτε ότι δεν είναι να κυβερνηθούν οι χώρες εκείνες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία δηλώσατε. Παρακαλώ να εξηγήσετε αυτά τα οποία είπατε και να αποσύρετε αυτές τις δηλώσεις γιατί ε, πήγεται η διαχείρισή σας ε, του κοινωνικού προπολογισμού και μιλούμε και για τους πόρους που από αυτές τις χώρες. Επίτροπος. Θεωρώ πως ε, στα κράτη-μέλη ε, υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα σταθερότητας. Αλλάζουν ε, κυβερνήσεις, έχουν ασταθεί σε κυβερνητικοί σχηματισμοί. Κυβερνήσεις που δεν έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών και δυνατότητα δράσης. Ε, σύντομα θα αποκτήσει μια κυβέρνηση που η Βουλγαρία που θα έχει την ικανότητα να δράσει όπως πρέπει. Ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευελιξία και τη μεταβίβαση επιστώσεων στα διαρθρωτικά ταμεία. Βάσει ε, της εμπειρίας μας ε, θα χρειαστεί όμως και προσπάθεια ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα. Ε, διότι υπάρχουν προγράμματα των διαρθωτικών ταμείων ε, που ε, υπάγονται σε εξαιρετικά περίπλοκες κατευθυντήρες γραμμές. Οπότε τα κράτη θα πρέπει να ενισχύσουν τη διοίκησή τους και σε συνεργασία με υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ούτως ώστε να υπάρξει τεχνική αρρωγή, τεχνική υποστήριξη προ τη δημόσια διοίκηση των κρατών με λόγια διαχείριση των προγραμμάτων. Και μπορώ να σα πω πως ε, θα χρειαστούν για πολλά χρόνια ακόμη τα προγράμματα των διαθροτικών ταμείων, διότι οι περιοχές τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται αυτά τα προγράμματα. Είμαι από τη Γερμανία και μπορώ να σα πω ότι μετά την ενοποίηση ε, το 89 δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν τα ανατολικά, πρώην κρατήδια ε, χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δευτερόλεπτα εκατομμύρια για την υποστήριξη των αδύναμων περιοχών. Ευχαριστούμε, ο Ρέμερ Μπέγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Σωστά είπατε ότι είναι ότι είναι βασική εξουσία αυτή που έχει το Κοινοβούλιο στα θέματα προϋπολογισμού και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, με αυτό το νέο γαλαξία και ε, ε μήπως ε, τελικά ο προϋπολογισμός θα ανατεθεί εξωτερικά, τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις για την παράταση του ΕΦΣΥ. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Και δεύτερον, ξέρετε ότι υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλία η οποία ακόμη συζητείται στην ε, ΕΚΟΝ και στην Επιτροπή Προπολογισμών για την ε, νέα δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνη. Ε, Πώ βλέπετε αυτό το ζήτημα, Είναι δυνατόν να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη αν δεν συμμετάχουν συμμετάσχουν ε, και τα άλλα κράτη-μέλη και πώς θα συνδυαστεί αυτό με τις προτάσεις για την αναθεωρήση του πολιτικού ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Απάντηση. Έρχονται στιγμές, όπως έλεγα, ε, που ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν με ευφυή και αποτελεσματικό τρόπο νέα εργαλεία. Ε, υπάρχει ε, στάσιμο πληθωρισμός, εν μέρη ύφεση ή χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ΕΦΣΙ και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο προκάτοχός μου φρόντισε σύντομα να υλοποιηθούν τα νέα μέτρα. Χρειάζεται όμως εξυγίανση, διαρθρωτική για τον προϋπολογισμό και γι' αυτό χρειάζεται να θεώρηση του του δημοσιονομικού πλαισίου και όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας, χρειάζονται αλλαγέ. Ε, τα ε, νέα εργαλεία όμως θα πρέπει να ενσωματωθούν μεσοπρόθεσμα στον προϋπολογισμό. Ε, εγώ πιστεύω ότι είχε καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμή ε, το ΕΦΣΥ. Την βασική αρμοδιότητα έχει ο αντιπρόεδρος Κατάινεν και ε, προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποια κράτη-μέλη μπόρεσαν να υλοποιηθούν ακόμη και νωρίτερα κάποια προγράμματα, χάρη στο ΕΦΣΥ και τη μόχλευση των κονδυλίων. Αυτή η βασική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου φυσικά αναγνωρίζεται. 26 ε, χρόνια ε, ήμουν ε, βουλευτής και Φυσικά αναγνωρίζω τη σημασία του Κοινοβουλίου. Θα είμαι πάντοτε ο εταίρος σας, διότι έχετε κάθε δικαίωμα. Πάντοτε θα υποστηρίζω το ρόλο του συνομοθέτη του Κοινοβουλίου για την διαμόρφωση των μελλοντικών πηγών εσόδων και των εξόδων του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστούμε. Καρτιά Ζαμπαλούδα. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνούμε ότι η Τράπεζα Επενδύσεων είναι βασικό παράγον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο ένα και περισσότερο συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έχουμε το πρόγραμμα Juncker, έχουμε και τις νέες τις ε, λοιπές αρμοδιότητες. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ανακτήσει ένα τμήμα αυτής της διαχείρισης που ανατέθηκε στην ΕΤΕ και για αυτό και είπατε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η, ε, η εντολή που της δόθηκε για το Ταμείο Εγγύησης, όπως επίσης και το πρόγραμμα για την Αφρική. Και το Συμβούλιο είπε όχι, πήγαμε σε διαπραγματεύσεις και εμείς, αλλά πέστε μας εσείς κύριε Τινγκερ, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει όσον αφορά αυτού την ανάκτηση της διαχείρισης του Ταμείου Εγγύσεων. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει μάχη για αυτή την ε, πρόταση έναντι του Συμβουλίου. Έτιγκερ. Ε, Πολύ συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων από τις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπής ε, και όλοι συμφωνούμε ότι ε, για ε, τα τραπεζικά καθήκοντα ενδείκνεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αξιολόγηση βερεκιώτες ε, για τα δηλωθετικά προγράμματα για τις ε, επενδύσεις. Επίσης, έχει εμπειρία και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδιαίτερη εμπειρία συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή προγραμμάτων διαρθωτικού χαρακτήρα και αυτό ισχύει και για το ΕΦΣΥ και για άλλες λειτουργίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο ή μόνο η Ευρωπαϊκή η ΕΤΕ ή μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, είναι αλληλοσυμπληρουμενη η ρολη μας και συνεργαζόμαστε και ε, αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Η ΕΤΕ έχει την ευθύνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα, δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε 16-18 δις εγγυήσεων ε, για το σχέδιο Juncker και για αυτά, ε, επειδή εντάσσονται στον προϋπολογισμό, έχει πλήρη δικαιώματα το Κοινοβουλίο για το Δημοκρατικό του έλεγχο. Ε, Χρειάζεται διαλειτουργικότητα ε, και συλλογική ευθύνη. Ε, δηλαδή, η Επιτροπή στηρίζει το έργο της ΕΤΕ και αντίστροφα. Μόρεσαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Τίνγκερ, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστούμε για τι τόσο συγκεκριμένε σα απαντώσει και την ξεκάθαρη θέση που έχετε για κάποια θέματα σημαντικά και όσον αφορά του ιδίου πόρου και όσον αφορά το επόμενο πολιτέ πλαίσιο υπολογίζουμε σε εσά σαν ε, σύμμαχο και έτσι με διαφάνεια να λειτουργήσουν ε, εύρυθμα στα νομικά και το, το δικό σα μικρό και το δικό μα. Δύο ερωτήσει. Πρώτα πρώτα, είδαμε πώ εξελίχθηκαν τα χρηματοδοτικά μέσα τα τελευταία χρόνια και το ΕΦΣΙ που είναι βασικό μέσο ε, πολιτική για επενδύσει. Είδαμε όμω τι γίνεται με κάποια κράτη-μέλη στην Ένωση που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια χρηματοδοτικά μέσα λόγω της ε, εξέλιξης των αγορών σε αυτά τα κράτη-μέλη. Βουκα, Βουκουρέστη, Σόφια, εξαρτώνται από Παρίσι και Φραγκφούρτο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτές τις χώρες. Οπότε πώς λέτε την ισορροπία μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων και των επιδοτήσεων και ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές ε, εμείς θέλουμε ε, σαν πολιτική ομάδα να δοθεί ένα ειστήριο ε, interest στους νέους που κλείνουν τα 18. Ε, η κυρία Γεωργίευα ε, που, προηγήθηκε τέλο πάντων σε αυτό το χαρτοφυλάκιο είπε ότι θα κάνει πιλωτικό πρόγραμμα για να χαρίσουν εισιτήρια ε, Interrail σε όλους τους 18 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. λέτε. Η Επιτροπή και εξετάζουν αυτή τη στιγμή την χρήση εγγύσεων του ΕΦΣΥ για προγράμματα στα κράτη-μέλη και στις περιοχές. Πώς ε, δεν εξετάζουμε μόνο ε, το θέμα των μικρών προγραμμάτων. Ε, θέλουμε να εξετάσουμε το, το θέμα και από την πλευρά των μικρών τραπεζών. Τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν. Ε, ποιος πρέπει να έχει το βασικότερο ρόλο. Τα τα κράτη-μέλη ΕΤΕ. Και επειδή υπάρχουν διαρθρωτικές ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχει αποφασιστικό ρόλο η ΕΤΕ ε, για την αποτίμηση της κατάστασης. Ε, φυσικά όμως θα δράσουν και εθνικές τράπεζε. Εάν προκύψει τραπεζική ένωση, αν λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά, ε, σε περίπτωση που είναι ασθενής ε, ή συντηρητικό ε, τραπεζικός τομέα μιας χώρα, θα πρέπει εξωτερικά να προέρθει μια χρηματοδότηση, να χρησιμοποιούνται οι εγγυήσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εθνικέ ή τοπικέ ε, κυβερνήσει ε, μέσα από διάφορε δράσει, ενημερωτικέ καμπανίε ε, να προσφέρει τελικά την υποστήριξη προ τι επιχειρήσει και τα μικρά προγράμματα. Για το Interrail έχουμε το Erasmus ε, την ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι χρησιμοποιούν αυτή την ελευθερία και το βρίσκω καταπληκτικό, διότι ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το, τη δυνατότητα να μετακινηθούν με το τρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυση αυτού του εγχειρήματο, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να βαρύνει και να λειτουργήσει ει του έρασμου. Ευχαριστούμε του συναδέλφου τη Επιτροπή των Προεκολών για τι ερωτήσει του. Ευχαριστούμε και εσά, κύριε Επίτροπε, που δώσατε τι ε, απαντήσει. Και τώρα θα με διαχθεί στην Προεδρία η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια γιατί ήσασταν επακριβέστατο στο χρόνο σα. Έχουμε τον κύριο Σαουάρμα λοιπόν πρώτο, ο συντονιστή. Ευχαριστώ, τον κύριο Σαρβάμα. Αγαπητέ Επίτροπε, θα σας ρωτούσα για το συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής της αρχής που να τον προπολογισμό που πρέπει να προστατεύεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως ο κύριος Άσκου, ο κύριος ήδη το ερώτησε αυτό. Πάντως εγώ δεν νομίζω ότι μας απαντήσατε με τρόπο συγκεκριμένο για την ερώτηση αυτή και θα την υποβάλω εκ νέου. Ποια θα είναι τα πρώτα σας βήματα ούτως ώστε να προωθήσετε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, το να εφαρμόσετε την αρχή του προσανατολισμένου σε αποτελέσματα προπολισμού. Όσον αφορά αυτά τα δεδομένα για, τον κρατικό, για τις κρατικές αρχές, αυτό για το οποίο κάθε χρόνο παραπονιέται το ελληνικό συνέδριο ότι έχουμε τόσα πολλά σφάλματα. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν τι θα κάνετε ούτω ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος. Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα από το χώρο της ενέργειας. Με το Connecting Europe Facility και την συγχρηματοδότηση υπερσυνοριακών υποδομών για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια ή αντίστοιχα δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας με στόχο την ανανέωση των ε, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε 1,9 δις από το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έπρεπε λοιπόν ξεκινώντας να ορίσουμε ένα στόχο. Ο στόχος ήταν η σύνδεση όλων των ευρωπαϊκών κρατών ε, και ενσωμάτωσή τους στην αγορά ενέργειας για το φυσικό αέριο και ε, την ηλεκτρική ενέργεια. Για να μην ε, χρειάζεται να προμηθεύεται από ένα μόνο τρίτο κράτος, κράτος μάλιστα Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φυσικό του αέριο. Η διαφοροποίηση οδηγεί εν τέλει στην μείωση των τιμών. Η Εσθονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Πολωνία ακόμη έχουν μπορέσει να αξιοποιήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την, ε, την διαφοροποίηση των πόρων των ενεργειακών και αντίστοιχα καλύτερες τιμές. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν μονοπόλιο, και αυτό το καταφέραμε, μειώνεται και το, ο κίνδυνος ενός μποϊκότ και ο κίνδυνος των υψηλών τιμών. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε όλοι σε αυτά τα προγράμματα, ορίζοντα του στόχου μα, του στόχου που είναι στόχοι που αστερνίζεται και ο Ευρωπαίος. Να του προσδιορίσουμε, να του επιδιώξουμε και να προσμετρήσουμε το αποτέλεσμα με βάση αυτού του στόχου. Ήταν πιο ευρωπαϊκή λοιπόν, πιο οικονομική συγγνώμη, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την μονομερή κίνηση των 28 διαφορετικών κρατών, των 27 όταν ήταν ε, τότε. Και βέβαια αυτό πάντα με τη διαφάνεια, με την απλούστευση, με απλές γραμμές, με παροχή συμβουλών στα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε από κοινού την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Η κυρία Γιάννα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, κύριε Έτυγκερ, να αναφερθώ σε όλες αυτές τις ε, αρμοδιότητε αλλά και σε αυτά που έχουν σχέση με τη χώρα σας. Έχετε τώρα αναλάβει τον προπολογισμό, αλλά και τις διαπραγματεύσει για τους επόμενου προπολογισμού. Εδώ και έξι μήνες όπως ξέρετε ε, επέμενε η Ισπανία για το θέμα των προστήμων που επιβάλλονται ει βάρος Πορτογαλίας και Ισπανίας. Ε, κάτι το οποίο σημαίνει πολλά εκατομμύρια από τα διευθυντικά ταμεία ε, και οπότε και οι δύο χώρες προέβησαν σε σημαντικές θυσίες. Επίσης οι άλλοι επίτροποι ήταν αποφασισμένοι να μην επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις. Εσείς όμως εμείνατε όλα αυτά δημοσιεύθηκαν στο γερμανικό τύπο. Οπότε και σας ερωτώ από πλευρά τη Ισπανία, εγώ ω Ευρωβουλευτή από την Ισπανία. Ανησυχώ για την αντίδρασή σα ει βάρο των ε, Ισπανών τόσα πολλά υποφέραμε και δεν μας βοηθήσατε. Εσείς επομένως, τι θα κάνετε εάν κάτι παρόμοιο συμβεί. Θα ξανακάνετε εσείς τα ίδια. Τι επιχειρήματα έχετε. Επίτροπο έχετε το λόγο. Στο θέμα της νοσομικής πολιτικής των κρατών. Πρέπει νομίζω ιδιαίτερα να μεριμνούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να μην διχαστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι έχει την αρμοδιότητα για την ε, εσωτερική αγορά, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ε, πάντοτε βλέπουμε να βάλετε με πολύ σκληρή κριτική. Έχω και εγώ ως επίτροπος δεχθεί κριτική ε, επικρίσεις από την Ισπανία, την Πορτογαλία και αντίστοιχα ή μάλλον αντίστροφα επιχειρήματα ήταν η πηγή των επικρίσεων από τη Γερμανία, τη Φιλανδία ή άλλα κράτη. Ο Επίτροπος, η δουλειά του είναι να αποφεύγει κάθε τι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διχασμό, σε διέρεση. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να τηρούνται οι κανόνε το six pack, το two το Maastricht. Αυτά δεν μπορούν να, ε, αλλάζουν κατά περίπτωση. Ε, Ρώτησε νωρίτερα ένας άλλος ε, βουλευτής εάν πάντοτε ισχύουν οι κανόνες, μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και βεβαίως έχω κάθε σεβασμό για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σας. Η σημασία των διαφορετικών προγραμμάτων όπως κράτη, για κράτη όπως Πορτογαλία, Ισπανία αλλά και τα νέα, νεότερα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ μεγάλες και τις γνωρίζω. Χωρίς ευρωπαϊκά προγράμματα πολλά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δηλαδή στα κράτη αυτά. Και γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της, Ευρωπαϊκής, της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος. Ναι, έχω γεννηθεί στη Γερμανία, ε, η καταγωγή μου είναι από τη Γερμανία, αλλά έχω ευθύνη απέναντι σε όλα τα κράτη-μέλη ως Επίτροπος και σε αυτό καμία, ε, η Γερμανία δεν έχει κανένα ρόλο. Τσαρνέτσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ισχύ σας Πρόεδρε. Έχω να σας υποβάλω μία ερώτηση. Έχουμε μία μελέτη κάποιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και για τον τρόπο που γίνονται αυτά συμφωνούν πάρα πολύ και άλλοι εμπλεκόμενοι όσον αφορά τα δεδομένα του FTS. Πώς μπορεί αυτό το σύστημα να βελτιωθεί και με τι χρονικό πλαίσιο. Επίτροπε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι κομμάτι τη κοινωνία των πολιτών είναι κομμάτι των δεσμεύσεων, των εθελοντικών, των εθελοντών, της προσφοράς στην κοινωνία. Συμπληρώνουν τη δουλειά του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής. Είχα λοιπόν ανέκαθεν αλλά και στα καθήκοντά μου τα προηγούμενα σε επίπεδο τοπικό, δημοτικό αλλά και μετά ε, μέγα σεβασμό για τη δουλειά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η υποστήριξή τους από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αντίστροφα, κάθε πρόγραμμα υποστήριξης θα πρέπει, ανεξαρτήτως του αποδέκτη των κονδυλίων, να καλύπτεται ε, να επαληθεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να γίνεται ο έλεγχο δηλαδή των λογαριασμών, να ελέγχεται και από το ελεγκτικό συνέδριο, να ελέγχεται από την Όλαφ, δηλαδή να ε, πράττουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μα ώστε να αποφεύγουμε ε, λάθη, ε, ακόμη και απάτη. Εδώ λοιπόν δεν θα παραλείψουμε τίποτα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η μειορθητήρηση δηλαδή, των ε, δημοσιονομικών κανόνων. Θα τηρούμε εμεί με απόλυτο τρόπο και απόλυτο σεβασμό του ε, δημοσιονομικού κανόνε, χωρί βέβαια να ε, εφαρμόζονται διακρίσεις εις βάρος ουδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάλλη, ευχαριστώ Επίτροπε και κύριε Πρόεδρε. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει των κρατών μελών στα πλαίσια της εξοπλίσης των κοινωνικών πόρων είναι η απλούσταυση. Έχουμε αυτή την πρότασή σας για το πώς να μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Άρα αυτό θα πρέπει και να γίνει, καλύτερη διοίκηση. Και έχουμε τώρα σημαντική περίοδο όσον αφορά το δημοσιογραφικό πλαίσιο. Άρα θα πρέπει όλα αυτά τα συστήματα να ε, επιληθούν. Εσείς θα συνεχίσετε αυτά το οποίο έχει υποσχεθεί να κάνει η προκάτοχό σας. και θα πρέπει να συνιστούν επομένω οι σχετικέ ε, προσπάθειε. Είναι απαραίτητο αυτό, ούτω ώστε να έχει περισσότερη αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και όσον αφορά τι επενδύσει στην Ευρώπη για το σχετικό ε, πλάνο. Οπότε το πλάνο Γιούγκερ μα θα πρέπει να υλοποιηθεί εσείς. Τι πιστεύετε για το ότι θα πρέπει τώρα να έχουμε πάρα πολλά ε, projects σε κράτη-μέλη τα οποία θα ωφεληθούν. Επίσης, επίσης την προσοχή σας σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση με το πρόγραμμα υλοποίησης του πολιτού πλαισίου. Για την περίοδο προγραμματισμού, εκεί οι πιστώσεις για το 2017 είναι πάρα πολύ περιορισμένες και αναβλήθηκε η ενίσχυσή τους. Οπότε εσείς τι συνέπειες βλέπετε ότι θα υπάρξουν για τον προϋπολογισμό και κυρίως εν ώψη και του Brexit. Επίτροπος. Σε όλα τα προγράμματα υποστήριξη κάθε επίπεδο πρέπει πάντοτε να διαφυλάσσουμε την ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης, της ε, μείωσης της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, της απλής χρήσης αφενός αλλά αφετέρου και την, της δίκαιης χρήσης, της αποφυγής ε, ανισορροπιών και ούτω καθεξής. Αυτό πάντα ισχύει, αλλά ισχύει ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε προγράμματα που ε, προσφέρουν υποστήριξη τοπικό επίπεδο, ε, όπως σε παραδείγματι στη δική μου την ε, κοινότητα για την ε, ανάπτυξη της απασχόλησης των νέων σε τοπικό επίπεδο, έχουμε διαφορετικά δεδομένα κάθε φορά. Έχουμε ακόμα και διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης ανάλογα με το κράτος μέλος και την περιοχή. Πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, ξέρετε, πάντοτε οι γεωργοί μου έλεγαν ότι ήταν πολύ περίπλοκο να ζητήσουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγαν ο Γεωργός ότι η δουλειά του είναι να πάει στο χωράφι, να φυλάξει τα ζώα του, να τα πουλήσει και το καθεξής και δεν θέλει να ασχολείται με την γραφειοκρατία. Ναι, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά ε, διαφορετικά προγράμματα για τη γεωργία, υπάρχουν τα προγράμματα για το greening, υπάρχουν ε, οι προτάσεις για την εκτακτικοποίηση. Ε, όλα αυτά περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τον Γεωργό και πάντοτε βρισκόμαστε σε ένα σπαγκάτ θα λέγαμε, σε μια δελκυστίνδα. Αφενός μεν προσπαθούμε με δεδομένη την εμπειρία που έχουμε από το, προ... από το πολιτισμικό πλαίσιο την προσπάθεια να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα εν ώψη του προσεχούς ε, κοιτάμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές απάτες ε, με ορθή διαχείριση και το καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτροπή, μία από τις ερωτήσεις αφορούσε το τι θα κάνετε με τα λόμπι. Ήδη κάναμε έξι συναντήσεις, πάρα πολλοί ήταν λομπίστες ε, που ήρθαν εκεί από μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις. Επίσης είχαμε και συνδικαλιστές και τα μικρή συμμετοχή άλλων εμπλεγωμένων. Μας είπατε τώρα ότι θα καλύψετε τα αιτήματα των μη κυβερνητικών Όμως, το πρόβλημα που συχνά ανακύπτει είναι ότι οι πόροι των λόμπι είναι πολύ περισσότεροι από τους πόρους που λαμβάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά πώς θα καλύψει τους λατές τις ομάδες των ενδιαφερομένων. Υπήρχε και κάποια ομάδα μοιραγωνομόνων που απεφάνθη ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου ε, αντιστάθμιση και αποζημίωση των εξόδων. Τι λέτε. τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλές ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με κυβερνητικές οργανώσεις, επέδο ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό. Και νομίζω ότι βλέπουν την ανάγκη για μια σταθερή χρηματοδότηση ε, προβλήματα ως προς το ύψο τη χρηματοδότησης δεν είχαμε ποτέ σε αυτές τις συνομιλίες. Αλλά πιο συγκεκριμένα, αν μιλήσουμε για το θέμα της ψηφιακή οικονομίας, υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα που είχαν διατυπωθεί από μικρές μεσές επιχειρήσεις, από ε, συνδικάτα, οργανώσεις εργαζομένων, εργοδότες, ε, βιομηχανία. Γιατί, ξέρετε, πολλές είναι χώρες που έχουν ιδιαίτερα δώσει έμφαση στην ψηφιοποίηση της κοινωνίας και δι για τις μικρομεσαίες, όχι για τη μεγάλη βιομηχανία τόσο. Και είχα την ευκαιρία πολλές φορές να επισκεφθώ χώρες ε, και περιοχές για να ενημερώσω για την ψηφιακή επανάσταση της μικρομεσαίας επιχειρήσης και τους επιχειρηματίες ε, βρισκόμαστε σε μια φάση όντω επανάσταση ψηφιακή. αν δεν προσέξουμε, αν δεν δώσουμε αρκετή προσοχή, κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο σε σχέση με τι ΗΠΑ και του ανταγωνιστέ μα στην Ασία. Και εδώ δεν μιλούμε για θέσει εργασία στην ε, βιομηχανία. Μιλούμε για θέσει εργασία για του νέου μα, για την επόμενη γενιά σε μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτέ τι εργασίε δεν τι δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί υποστηρίζουμε βεβαίω με κάποια ποσοστά και στόχου που ορίζουμε, αλλά τι θέσει εργασία θα τι ε, δημιουργήσει ο επενδυτή. Ε, οι υποδομέ που θα δημιουργηθούν. Και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να δεχτείτε αυτό που σας λέω ότι κάνω ό,τι μπορώ στις συνομιλίες μου με τους εκπροσώπους των φορέων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για την διαφύλαξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Και όχι μόνο με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συνομιλώ και με τη Huawei, την Alibaba, την, ε, ε, την ε, Hewlett Packard, οτιδήποτε μπορώ να κάνω ώστε να ενισχύσω την ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά, ανεξαρτήτως κομματικής προελευση κάθε υπουργό. Ε, Ανάπτυξη. Ε, φιλελεύθερος είναι χριστιανοδημοκράτη, είναι πράσινος, στη Γερμανία έχουμε και πολλού πράσινους. Κάνει το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή προσπαθεί να βελτιώσει την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου ψηφιακής οικονομίας, ως κέντρο της ψηφιακής οικονομίας. Παρακαλώ. Ο κ. Γεύρο, από το 2014 έχετε δει πολύ περισσότερο τους εκπροσώπους της παρά όλους τους άλλους εμπλεκομένους στις αρμοδιότητες σας. Και ήταν πάρα πολύ περί αυτά τα οποία είπατε όσον αφορά εκείνη την ε, μετακίνησή σας με το αεροπλάνο. Και είναι και το θέμα των λόμπι. Άρα η προσωπική σας προϊστορία με τίποτα δεν μας εγγυάται τη τήρηση των όσων έχετε υποσχεθεί για τη διαφάνεια. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη. Τι συγκεκριμένα θα κάνετε ούτως ώστε να κάνετε πιο άρτιο τον κονισμό για τα λόμπι, αλλάξετε αυτούς τους ισχύοντες κανόνες. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι στο μέλλον θα επιβληθούν οι κυρώσεις εκεί που πρέπει σε σχέση με τις αρμοδιότητές σας. Κύριε Βουλευτά, θα ήθελα για την προσωπική μου προϊστορία ε, να μιλήσετε με τον Ρέινχαρντ Μπιούτεκόφερ. Ε, γνωρίζει τις αδυναμίες μου και έχω αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι προκατηλημένος και μπορεί να λειτουργήσει ως αμερόληπτος δικαστής ε, διότι με γνωρίζει από το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι σε θέση να αξιολογήσει τις προηγούμενες επιδόσεις μου. Βασικό σημείο για το οποίο αγωνίστηκα ήταν η ψηφιακή επανάσταση, η ευρυζωνικά δίκτυα, ε, οι τηλεπικοινωνίες. Είναι βασικός τομέας, δεν είναι οποιοδήποτε τομέας. Η ψηφιακή υποδομή της Ευρώπης δεν είναι καλή. Πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία των Megabit. Χρειαζόμαστε λοιπόν την οικονομία των τηλεπικοινωνιών. Όλες όλες τις επιχειρήσεις, οι Ευρωπαίοι παίκτες ε, οι εθνικοί, οι περιφερειακοί και οι τοπικοί παίκτες πρέπει να συμμετάσχουν και οι Και γι' αυτό ε, συναντήθηκα ε, τακτικά με εκπροσώπους ενώσεων ε, για την ε, οδηγία ETS, ETMS που μετά τον τριμερή διάλογο αποφασίστηκε και έτσι σχεδιάσαμε το τηλεπικοινωνιακό πακέτο. Το Σεπτέμβρη, πέρσι, καταλήξαμε ε, σε συμφωνία ε, για αυτό το τόσο σημαντικό πακέτο. Και καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω την τεχνογνωσία του κλάδου. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι το ρόλο που καλούμε να διαδραματίσω. Για την ε, ψηφιοποίηση της οικονομίας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια επενδύσεων ε, για τα, τα 5G, για τις οπτικές σύνδεσεις χρειάζονται 500 δις επενδύσεις. Δεν γίνονται αυτά χωρίς τον κλάδο. Γι' αυτό για συναντήθηκα με τις ενώσεις εκπροσώπους τους επιχειρήσεις και ε, δεν βλέπω για ποιο λόγο ε, θα ήταν επιλήψιμο αυτό. Έτσι αντιλαμβάνομαι το ρόλο του Επιτρόπου για αυτή την οικονομία. Ευχαριστούμε. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα διότι ο συνολικός χρόνος είναι τρία λεπτά. Ε, η FTD βάλει... δεν τον βλέπω τον κύριο Βάλη. Ποιος θέλει, να, κάποιος να πάρει τη θέση του. Όχι. Σταϊχόφσκι τότε. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι η ερώτησή μου θα σας ενοχλήσει τόσο όσο οι ερωτήσει των άλλων συναδέλφων. Εργάζομαι στην Επιτροπή Λέχων Προπολογισμού και θα σα ρωτήσω το εξή. Κάποια θεσμικά όργανα δεν είναι πρόθυμα να συνεργαστούν όσον αφορά του οικονομικού ελέγχου και όσον αφορά τη διαδικασία για τι ε, απαλλαγέ. Φερρυπίν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αποφεύγει εδώ και πολύ καιρό τι ε, συζητήσει για του οικονομικού ελέγχου επί των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους Ευρωπαίους. Να, δεν υπάρχει διαφάνεια στα θεσμικά οργάνα, λέει ο κόσμος. Εσείς τι θα κάνετε για αυτό το πρόβλημα. Το γνωρίζετε το πρόβλημα. Τι θα κάνετε. Και ε, μια άλλη σύντομη δεύτερη ερώτηση, συμπληρωματικά στα όσα είπαν οι συνάδελφοι που με ε, εκάλυψαν καταρχήν, για το τι θα γίνει το 2020. και για την περίοδο 2021-2028. Ε, Θα καλύψετε τις νέες προτεραιότητες για την ιστορική ασφάλεια και την καινοτομία σε εκείνους τους κύριε Βουλευτά. Ναι, αμφισβήτητα. Φυσικά η ε, δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες και τους υπαλλήλους ε, της δημόσιας διοίκησης. Είτε μιλάμε για το Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο ε, των Υπουργών, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να αλλιώς να εργαστούμε με σταθερό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αποδοχή, έτσι λειτουργεί η δημοκρατική ε, κοινωνία. Ε, ανεξαρτήτως για ποιον μιλάμε. Και σίγουρα σε αυτό, επιδέχεται βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πού μπορεί να βελτιωθεί στην επικοινωνιακή της πολιτική, στα ΜΜΕ, τα κοινωνικά μίντια, ε, στις ε, διασκέψεις, στην παρουσία της ε, εκτός Βρυξελών στις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι εσείς, επειδή έχετε τις εκλογικές περιφέρειες σας, επειδή έτσι είναι ο ρόλος σας, ε, δεν ε, ε, μπορούμε να παραναβελτιωθούμε και χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με άλλους τομείς. Κανείς η υπουργό δεν λειτουργεί με τόσο διαφανή τρόπο όπως εμείς. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ένας βουλευτής εκπροσωπεί πάρα πολλούς πολίτες και το ίδιο ισχύει και για τους επιτρόπους, η αντιστοιχία δηλαδή ανάμεσα στον αριθμό των πολιτών και τον αριθμό μας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο, να ενημερώνουμε για τη δουλειά μας. Για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο Είμαι βαθύτατα απεπισμένος ότι στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας υπάρχει προσθέμενη αξία από πλευράς της Ευρώπης και τους επόμενους, ε, το, ε, τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η προσθεμένη αξία, το αντίθετο. Ευχαριστούμε Γκάιερ. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών υπάρχουν ε, σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με το ποσοστό λαθών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Πώς μπορεί να μειωθούν αυτά τα λάθη. Ε, δεν χρειάζεται τώρα να πω σε λεπτομέρειες νομίζω. Το θέμα ε, είναι η νομοποίηση ίδια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η μείωση του ποσοστό των λαδών θα έχει αποφασιστικό ρόλο και γνωρίζετε ότι ακόμη και για τις ακροδεξιές δυνάμεις μπορούν να, μπορεί να υπάρχει κατάχρηση ακόμη και τυπικών λαθών, ε, διότι το εξισώνουν με απάτη και διασπάθηση του χρήματος. Ε, πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε από κοινά πώς μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό των λαθών. Για την εκτέλεση του προπολογισμού υπάρχουν τομεί όπω η ανάπτυξη τη υπέδρου και η περιφερειακή πολιτική, όπου ε, κατά παράδοση είναι ιδιαίτερα υψηλά ποσοστό των λαθών. Και ε, το ελεγκτικό συνέδριο κάθε χρόνο το τονίζει, διότι τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, μπορούν να διορθώσουν τα λάθη λόγω και έλλειψης ε, πληροφοριών, ε, έλλειψης δεδομένων. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω, εσείς τι προτείνετε να κάνετε ακριβώς για τη μείωση του ποσοστού λαθών. Απάντηση. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το τομέα και ενημερώθηκα τις τελευταίες εβδομάδες γι' αυτό. Έχω συλλέξει πάρα πολλέ πληροφορίες και μπορώ να σας πω ότι αυτό που πρέπει να κάνετε είναι ακριβώ να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Δεύτερον, το ποσοστό λαθών τουλάχιστον ακολουθεί ενάρετη πορεία. Ε, έχουμε φτάσει στο 3,8 από το 5,4. Η ανάκτηση των ε, ποσών μετά την, ε, τον εντοπισμό των λαθών ε, ακολουθεί επίσης θετικό προσανατολισμό, οπότε δεν μπορούμε να το εξισώνουμε με απάτη. Λάθη, γίνονται τα λάθη, είναι ανθρώπινα. Το θέμα είναι η διόρθωση των λαθών, η ανάκτηση των ποσών και η περαιτέρω μείωση του ποσοστού των λαθών. Να πέσουμε κάτω από το 2%. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και ε, πώς θα συνεχίσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο. Άρχισε επαφές με τον νέο πρόεδρο και η πολιτική για τη μείωση των λαθών ναι, συνδυάζεται με την πολιτική για την βελτιωμένη αποδοτικότητα και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με την αποδοχή των πολιτών για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούμε σωστό δρόμο. ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίση είναι στοχευμένη κίνηση και θα συνεχίσω τον δρόμο που χάραξε η κυρία Γεωργίευα. Δηλαδή, ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια προ όφελο του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Όλο αυτό το οπλοστάσιο θα μας βοηθήσει και κατά τη δική μου αποτίμηση ε, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην γεωργική πολιτική από στη διαρθρωτική πολιτική. Ο κύριος ε, Τσερνεύσκη έχει παραχωρήσει το χρόνο μιλές ομάδος του. Καλή χρονιά πρώτα πρώτα κύριε Επίτροπε. Βλέπω ότι είναι καλή η διάθεση των συναδελφών κάνουν πλάκα. Λένε το ανέκδοτο. Το ότι τα λέτε πολύ συγκεκριμένα, συγκεκριμένε απαντήσεις, αλλά εγώ δεν διαπιστώνω κάτι τέτοιο. Κάτι που ενδιαφέρει την Επιτροπή Προπολογισμού. Μας είπατε στις ε, απαντήσεις ότι θέλετε τον προπολογισμό που να στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και είπατε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο και ότι στο μέλλον επίσης θα υπάρξει επίπτωση στον προπολογισμό και σε όλους τους ε, εμπλεκομένους. Όμως, λείπουν δύο πάρα πολύ βασικά στοιχεία. Τι γίνεται με την ε, πρωτοβουλία, τον ηγετικό ρόλο, αυτό το leadership του προπολογισμού αποτελεσμάτων. Πού είναι αυτό το leadership, ποιος θα είναι αυτός ο βασικός ε, παράγων ή σύμβουλος για τον προπολογισμό. Πώς θα εξασφαλίζεται τη συνέχιση της διαδρομής της προκατόχου σας. Τι συγκεκριμένα θα κάνετε. Και κάτι άλλο. Ο συνάδελφος πριν ανέφερε για την πτή σας με το ιδιωτικό jet. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες η χρήση τέτοιων ιδιωτικών jet. Άρα, κομμένη πλάκα και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Επίτροπο. Zum zweiten Punkt habe ich Έχω δώσει πλήρη αιτιολόγηση, ε, διότι, ξέρετε, έχω απαντήσει στη γραπτή σας ερώτηση ε, για αυτό το θέμα. Ας αρχίσουμε όμως με τον προπολογισμό επί τη βάση αποτελεσμάτων. Ε, θα πρέπει τομεακά να κινηθούμε. Ξέρουμε, παραδείγματο χάρη στον ενεργειακό τομέα, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ε, μονοπόλια, υπάρχουν προβλήματα ε, εφοδιασμού. Ε, ανέφερα τι βαλτικέ χώρε. Και μετά μιλάμε για αποτελέσματα. Δηλαδή να έχουν περισσότερους προμηθευτές, περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερους αγωγούς, περισσότερη δυνατότητα αποθήκευσης. Γι' αυτό κράτη-μέλη όπως η Λιθουανία, η Φιλανδία, η Εστονία, ε, η Λετωνία χρειάζονται χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε εμείς ότι ο στόχος θα πρέπει ε, να είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας ε, και στον τομέα του φυσικού αερίου θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτό πώς θα γίνει όμως με διασύνδεση των αγωγών. Χρειαζόμαστε τερματικούς σταθμούς LNG να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης και να αποτεμήσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής μειώθηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Υπάρχουν περισσότεροι προμηθευτές, έχουμε περισσότερες πηγές, περισσότερη αγωγή. Ναι ή όχι και να δούμε αν ήταν επιτυχημένα τελικά τα προγράμματα νέου. Ναι, και αυτή η leadership, αυτός ο ε, ηγετικό ρόλος που είπατε, πέρα από του βασικού επιτρόπου υπάρχουν και οι ε, κατατομία αρμόδιοι επιτροποί για τις ε, επιδοτήσεις ανατομέα, για την υποδομή, για την προώθηση της απασχόλησης, για τον πολιτισμό και το καθεξής. Λοιπόν, και υπάρχει και ο, ε, ο ρόλος του καθενός. Ε, ελέγχουμε τους εαυτούς μας ε, και βλέπουμε ότι ε, χρειαζόμαστε στοχοθέτηση, η οποία δεν προέρχεται όμως αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, θα πρέπει στις υποσημειώσεις να βλέπουμε την αιτιολόγηση για κάθε στόχο, γιατί εσείς δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτούς τους στόχους με την έγκριση του προπολογισμού. Και λοιπόν, να, λέμε, να διαπιστώνουμε αν σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι. Μαζί θα, θα έχουμε αυτό τον ηγετικό ρόλο και μαζί θα κάνουμε και την αποτίμηση. Αυτή ήταν η ιδέα τη ε, κυρία ε, Γεωργία. Ναι, ευχαριστούμε διακόπτη κυρία Γκρέσλη. Για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει με συνέπεια αυτή την οδρο αυτή την οδό να ακολουθήσουμε. Ashworth από το ECR. Επίτροπε, βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των ψήφων κατά του κατεστημένου ε, Πάρα πολλοί είναι τώρα οι Ευρωπαίοι που τη βλέπουν μακρινή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βλέπουν πάρα πολύ γραφειοκρατική, που πιστεύουν ότι δεν δουλεύει για το καλό τους. Και όλοι οι ευρωσκεπτικιστές έχουν τα πιο ισχυρά επιχειρήματα με τον προπολογισμό. Μπορείτε να επηρεάσετε πάρα πολύ την εξέλιξη ούτως ώστε να ξανακερδίσουμε τους Ευρωπαίους. Πώς μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, λέτε. Ε, να προωθήσουμε, να διαφημίσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Ναι, ε, ξέρετε ότι προβλέπονται κονδύλια γι' αυτό, ε, Προβλέπετε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ε, πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα όπου με πιο αποτελεσματικό τρόπο μπορούμε να έχουμε τα επιδιακόμενα αποτελέσματα. Στον τομέα της έρευνας, παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα για το High Performance Computing. Ε, τη δεκαετία του 80, από τις 10 δυνατότερες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό ε, ήταν στην Ευρώπη. Τώρα όμως ε, έχει μείνει μόνο μία. Δεν χρειαζόμαστε όμως υπερυπολογιστές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε δύο-τρεις που θα είναι στη διάθεσή μας για ερευνητικούς στόχους, για τον κλάδο της έρευνας. Χρειαζόμαστε κοινή προσπάθεια και γι' αυτό έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια να συγχρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα με εθνικά μέσα, να έχουμε δύο-τρεις σούπερ ε, ε, στην Ευρώπη ε, και μόνο έτσι θα έχουμε αποτελεσματικότητα στις επενδύσεις. Και μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα σε άλλους τομείς όπου φυσικά θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει σεβαστή και η αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να υπάρχει λόγος για την ευρωπαϊκή παρέμβαση αποτελεσματικότητα, αλληλεγγύη. Αυτοί είναι λόγοι. Ε, ή ε, επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε Αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να νομιμοποιείται η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε ευρώ που εκταμιεύουμε θα πρέπει να αναφέρουμε για ποιο λόγο το κάνουμε. Δικαιολογούμε ε, στα μάτια των φορολογουμένων. Για, αυτό το, για ποιο λόγο πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο να δραστηριοποιηθούμε. Η κυρία Σμίτ. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Μου στείλατε απάντηση για τα μελλοντικά προγράμματα ε, που έχετε για το Ευρωπαϊκό Ναυτοεξιακό Ταμείο και ε, την ένταξή του στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα το 2020. Είπατε ότι θα ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα και θέλω να ρωτήσω, δεν εξυπηρετεί το στόχο μας ε, καλύτερα να εντατικοποιήσουμε τώρα τις συζητήσεις μας και να κάνουμε μια πιο ευέλικτη παρέμβαση στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ναυσιακού Ταμείου και επίσης σε σχέση με τον Brexit ε, και των υπολοιπόμενων κονδυλίων δεν θα πρέπει ε, να ε, στοχθετήσουμε καλύτερα τη χρηματοδότηση που προβλέπουμε για το επόμενο πολιετές πλαίσιο και μήπως χρειάζεται στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Ναυτοξιακού Ταμείου με αποτελεσματικό τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει καλύτερο συντονισμό, δηλαδή απάντηση. Ναι. Ευελιξία χρειαζόμαστε ανάμεσα στα προγράμματα ε, και στους τίτλους αλλά και στα ε, έτη, τα οικονομικά έτη του προϋπολογισμού. Ε, και νομίζω ότι αυτό θα ε, το επιτύχουμε, θα διερευνήσω κάθε πιθανότητα που υπάρχει στην, ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιο. Υπάρχει η ε, διαφάνεια και η πραγματικότητα που ισχύει στον προπολογισμό. Έχουμε τόσα δισεκατομμύρια και προσπαθούμε με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ανάλογα με τι ανάγκε μα, να εκταμιεύουμε τα κονδύλια. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όμω, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ταυτόχρονα να παραμένουμε ευέλικτοι και νομίζω ότι αυτέ είναι σωστέ κατευθύνσει. Για το ε, αναπτυξιακό ταμείο, Ε, κοντεύει να κλείσει τα 60 χρόνια και έχει αυξανόμενη σημασία σε σχέση με το παρελθόν, διότι συνδυάζεται με την αναπτυξιακή μας πολιτική, την πολιτική γειτονία, ε, τη χρηματοδότηση προοπτικών ως προς την παιδεία, την ασφάλεια στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και των μεταναστών, διότι αυξάνεται το πρόβλημα, δεν μειώνεται. Ε, και γι' αυτό ε, στην ε, διάμεση αναθεώρηση του πολιετούς και στο επόμενο πολιετές θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως πρέπει να ενταχθεί ή να πλησιάσει τουλάχιστον τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και το ξαναλέω και το τονίζω. Ε, θα, καλύτερα είναι να έχουμε κονδύλια ε, εκτός παρά να μην έχουμε επαρκή κονδύλια εντός του προϋπολογισμού. Πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε το Συμβούλιο όμως. Πρέπει να παίξει μπάλα και το Συμβούλιο μαζί μας. Και ε, τα χρειαζόμαστε τα λεφτά που θα εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, για το Brexit. Να ξαναπώ Ευχαριστώ ότι είναι ένα έκτακτο γεγονός ε, το οποίο πρέπει θα να αντιπεξέλθουμε αλλά επί της αρχής πιστεύω ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να είναι, έχει αναδειχθεί μάλλον σε ε, ευρωπαϊκό καθήκον και γι' αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Σέλσος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ. Επιτροπή. Σήμερα με την επιστολή Γιούνκερ της πρώτης στην δεκάτω του 2014, πρέπει τώρα να είστε επικεφαλής της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του ε, δημοσιονομικού πλαισίου και επίσης για τους βγουν μετά το 2020 και έτσι να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα συστημικά προβλήματα του κοινωνικού προϋπολογισμού. Συμφωνίζετε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επάρκεια πόρων στον προπολογισμό. Θα αναλάβετε δράση σε σχέση και του ψηφίσματός μας του Ιουλίου του 16 εκεί τονίσαμε ότι οι οροφές του πλαισίου είναι πολύ ανεπαρκείς και εγώ το σύστημα τώρα έχει φτάσει στα ωριά του. Το ζωτομάτων μάλλον εφόσον ε, στην ίδια επιστολή είχε τονίσει ο πρόεδρος Γιούνκερ ότι σήμερα ζούμε σε κάποια ένωση που υπάρχει το 21ο κράτος μέλος. Οι άνεργοι, πολλοί εκ των οποίων είναι νέοι, αισθάνονται ότι έχουν περιοριοποιηθεί και οπότε θα πρέπει αυτή η άνοιγη να είναι το πρώτο μας μέλημα. Συμφωνείτε ότι η αυτών ε, το 1 δισεκατομμύριο για αυτή την πρωτοβουλία για τους νέους ανέργους. Δεν είναι φραγκοδίφραγκα. Και απαντήσατε στον κύριο Μάνκα ότι περιμένετε τι θα πει το Συμβούλιο και είπατε και στον κύριο Λεβαντός για τους ιδίους πόρους. Είπατε ότι η έκθεση Μόντι είναι απλά μια έκθεση. Δεν δεσμεύει. Ε, δεν συνάδουν με την ηγετική αποστολή σας για αυτά τα θέματα. Εάν το κανονιστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο δεν αποδίδει, τότε θα πρέπει να επανασχεδιαστεί. Δεν είμαστε business as usual. Ε, έχουμε μπουχτίσει. Απάντηση. Η Επιτροπή έχει κάνει από το προηγούμενο φθινόπωρο τη δουλειά της σε σχέση με τις προτάσεις και τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Τώρα πρέπει να πείσουμε την Ιταλική κυβέρνηση να συνεργαστεί σε μια απόφαση του Συμβουλίου και μετά θα είναι δική σας η σειρά για τι διαπραγματεύσει μεταξύ Συνοβουλίου και Κοινοβουλίου τις οποίε εγώ θα συνοδεύσω, θα δίνω ίσω ενάυσματα, προτάσει ιδέε. Έχουμε καταφέρει μερικά πράγματα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να προχωρήσουν αυτά τα, αυτές οι προτάσεις και ώστε να έχουμε επαρκείς πόρους για τις δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια, για την ανάληψη υποχρώσεων Η πρικοδότηση διαρθρωτικά και θα σας το πω πολύ απλά γιατί ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει πολύ εύστοχα επιχειρήματα ώστε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι αλλά ταυτόχρονα υπάρχει από την άλλη και το Συμβούλιο. Λοιπόν, εγώ θα παραμείνω σε όλη μου τη ζωή ένας ε, έντιμος διαμεσολαβητή, συνήγορος στο ΣΥΠΗΝ, για να προχωρήσουν οι προτάσεις αυτές. Για την απασχόληση των νέων, ένα πράγμα είναι οι εγγύησεις, άλλο πράγμα είναι το χρήμα που χρειάζομαι για να δώσω ευκαιρία για ένταξη στην αγορά εργασία στους νέους. Και θα το χρειαστώ για αρκετά χρόνια κατά πάσα πιθανότητα. Άρα θα χρειαστώ επαρκή πρικοδότηση και αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και Πρόεδρε. Υπάρχουν ακόμα Μεγάλε αδυναμίε ω προ την διαχείριση και του ε, ελέγχου σχετικού με τα διαρροτικά ταμεία. Γιατί έχουμε πάρα πολλέ ε, απάτες που δεν αναφέρονται από τι κρατικέ αρχέ, μα είπατε προηγουμένω, Επίτροπε, διαφορά μεταξύ σφάλματο και απάτη. Όμω, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι απώλειε είναι δισεκατομμύρια και προέρχονται από τις τσέπες των φορολογουμένων. Έχουμε παρατυπίες, έχουμε απάτε και οι σχετικέ καταγγελίε παίρνουν χρόνια για να διελευκανθούν. Θα πρέπει να υπάρξει επομένω κάποιο σύστημα fast track. Εσείς τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ούτω ώστε η έλεγχη και η διαχείριση να είναι όπως πρέπει ο πλευράς των κρατών μελών. Μήπως θα πρέπει να υπάρχουν ε, αυστηρότερες κυρώσεις στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο είδου απάτη ή παρατυπία. Και ε, στο παρελθόν ακαδημίλια αξιοποίησαν τα κοινωνικά κονδύλια και βελτιώσουν την οικονομία τους. Άρα θα πρέπει να γίνει πιο σοβαρός διάλογος με τα κράτη-μέλη που αξιοποίησαν έτσι τους πόρους και θα πρέπει επίσης να συνοηθούν εκείνες οι χώρες με τις χώρες μέλη που ακόμα πασχίζουν να κάνουν το ίδιο με βοήθεια τους κοινωνικούς πόρους. Δεν θα θέμα Επιτροπής, είναι θέμα κρατών μελών. Ο Επίτροπος. Οι εκθέσει που θα υποβάλω φέτος θα, θα δώσουν την έμφαση στην τη Όλαφ. Δεύτερον, στην ΕΠΟ βλέπετε την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ως εκ τούτου μια καλή ευκαιρία βλέπω εγώ να μην παρεμποδιστεί η σχετική εξέλιξη από το Συμβούλιο. Αρμοδιότητες σχετικές με, τους, με, τους, ε, με το φόρο είναι μια διεκδίκηση στην οποία συνεργαζόμαστε, θα αγωνιστώ και εγώ, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε συμπληρωματικά σχέση με τις εξελίξεις με τον Ηνωμένο Βασίλειο και την Όλαφ. Η ερώτηση σχετική με τα παλαιά έναντι των νέων κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος, πιστεύω, μπορεί να αντλήσει πλέον εκτήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορεί κάποια κράτη-μέλη να αντλούν πόρους, άλλα όμως κράτη θέλουν την εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει καμία περιφέρεια να μένει πιο αδύναμη. Να δώσω ένα παράδειγμα από την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Με τα διευθυντικά προγράμματα. Πηγαίνουν χρήματα στην Πολωνία. Αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και μεγάλα ευκαιρίε για οικοδομές, για εργαλεία, για εργαλειομηχανές, βαρέα μηχανήματα, φορτηγά, ξαφικά και το καθεξής που επανέρχονται στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προστεύουμε τόσο πολύ τα ωφέλη προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Όλοι μπορούν να υποφεληθούν, να ενισχυθούν όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης και μπορέσουν σιγά σιγά οι πιο αδύναμες ε, περιφέρειες να γίνουν πιο ισχυρέ στην Ευρώπη, να έρθουν πιο κοντά στι ισχυρέ. Κύριο Γκάιερ, ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι με τα τελευταία σας λόγια ε, αποδείξατε ότι δεν είμαι ο μόνος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει η έννοια του καθαρού εισφέροντος στον λογαριασμό. Είμαστε δύο, εσείς και εγώ δηλαδή δεν το έχουμε καταλάβει αυτό σαν έννοια. Βεβαίω και όλοι αντλούν πλέον εκτήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και οι πιο ισχυροί οικονομικά και οι λιγότερο. Ε, εδώ λοιπόν έχω να πω ότι με απασχολείται το θέμα των λόμπι. Δεν υπάρχουν συζητήσει είτε εδώ, είτε στις Βρυξέλλε, είτε οπουδήποτε στη Γερμανία που να μην βλέπουμε εμφανή το ρόλο των λόμπι, των ομάδων πιέσεως. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι λοιπόν στο ποιο μιλάει με ποιον. Αυτό το κάνουμε όχι για να χαλιναγωγήσουμε τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά για να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ έχω ανοιχτή την πόρτα σαλδημοκράτης στα συνδικάτα, στις κοινωνικές ενώσεις και την εκκλησία, την ε, ε, θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκω. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα, αλλά πρέπει να είναι και δημόσια ξεκάθαρο, για να μην υπάρχει επίδραση στις πολιτικές επιλογές ε, των πολιτικών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος πιστεύω ώστε να ε, διασκεδαστούν και οι επιφυλάξεις και οι υποψίες ακόμη του πολίτη έναντι της δουλειά μας. Πρέπει να είναι δημόσιο λοιπόν, δημόσιο κτήμα του ποιος μιλάει με ποιον. Πρώτη δήλωση και αξίωμα. Δεύτερον, λέτε ότι ε, μπορεί να επηρεαστεί κάποιος ακόμα και αν δεν ε, ορίζεται ξεκάθαρα. Ε, επί παραδείγματι κάποιες συναντήσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με κάποιους που δεν καλύπτονται στο μητρό των λόμπι. Αυτό το επιχείρημα δεν μπορώ να πω ότι το δέχομαι. Συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει στο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στο ποιο συνομιλεί με ποιον και ποιες ιδέες φτάνουν την Επιτροπή από κάποιους παράγοντες εκτός αυτής. Ο κύριος Έτεγκερ, για την πρώτη ερώτηση, ανεπιφύλακτα θα απαντήσω ναι. Για τη δεύτερη, είμαι ετεθειμένος μαζί σας να επαληθεύσουμε, να εξετάσουμε το τι είδους καταχώρηση μπορεί να είναι υποχρεωτική, με ποιοι όροι θα πρέπει να είναι αυτοί που θα οδηγούν στην καταχώρηση των Μητρό των λόμπι και να το δούμε αυτό σχέση και με τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Στην πατρίδα μας, τον Τίσελ, το Χάρδι το Βερολίνο, είναι αυτονόητο αυτό που λέτε, δεν το συστάει κανείς. Ε, υπάρχουν ιδέες λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις και μπορούμε τις γκρίζες ζώνες να τις απαλείψουμε τον τρόπο αυτόν. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα κάπως ασαφή. Εγώ, παραδείγματι, είμαι φίλος εδώ και χρόνια με έναν ε, επίσκοπο της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Ε, χρόνια τώρα, ε, τηλεφωνήματα, επαφές, ε, συνομιλίες, γενέθλια, χρόνια πολλά. Αυτό θα μου, το, θα μου πείτε ότι είναι λόμπι ή ότι είναι μια φιλική σχέση. Γιατί υπάρχουν πολλά αντίστοιχα τέτοια. Μπορεί να συναντήσω κάποιος σε ένα αεροδρόμιο. Να διαβάζω ε, ε, μου έχει συμβεί μάλιστα να διαβάζω εφημερίδα έτσι ψηλά πάνω από το κεφάλι μου στο αεροδρόμιο για να μην με αναγνωρίσει κανεί και έρθει να μου μιλήσει. Γιατί ε, και ένα κοινό πολίτη μπορεί να έρθει να με αναγνωρίσει και να μου ζητήσει κάτι. Πού θα βάλουμε το όριο λοιπόν για το λόμπι. Εγώ λοιπόν προκαλώ οποιονδήποτε και εσά στην πολιτική σα ομάδα ή σε οποιοδήποτε πολιτικό όργανο να μου δώσει συγκεκριμένου όρου απόλυτα σαφεί και ασφαλή για το πώ θα αποφύγουμε το λόμπι. Η κυρία Γκρέσλε. Ναι, θέλω και εγώ να πω δύο λόγια ε, σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης ως ομιλήτρια. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με την απάτη, νομικά ζητήματα, προτάσεις, ε, διατάξεις που βεβαίως στόχο έχουν να μην παρεμποδίσουν την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων, αλλά και να αποτρέψουν ταυτόχρονα τι απάτε. Πώ μπορείτε λοιπόν να οργανώσετε εσεί το επιτελείο σα, ώστε να σα βοηθεί το προσωπικό σα στην επιτέλεση του έργου σα, χωρί βέβαια τέτοιε επιρροέ, και αφετέρου για την αξιολόγηση. Μας λέτε ότι η αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα προκύψουν από τη δουλειά ενό Ινστιτούτου. Ποιο είναι αυτό και τι μπορούμε να περιμένουμε. Κύριο Σέτεγκερ, κοιτάξτε, δεν έχω υπόψη νομική βάση αυτή τη στιγμή που να με εμποδίσει να κοινοποιήσω στο Κοινοβούλιο τη σχετική έκθεση. Εάν δεν υπάρχει απαγορευτική διάταξη, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει αυτό να μην συμβεί. Πολύ ευχαριστώ να έχουμε τη σχετική επαφή, η Επιτροπή σας, τα μέλη του επιτελείου μου και βεβαίως ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στην καταπολέμηση της απάτης Πρόκειται για μια έκθεση λοιπόν που έχει ε, εκδοθεί από ένα ιστοτοπό που ασχολείται με την απάτη. Είναι μια, ε, ένας φορέας ο οποίος ασχολείται ειδικά με τα θέματα αυτά. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα μου είναι χρήσιμη σε όλη μου την ε, πορεία και θα την λάβω υπόψη μου σε όλες μου τις δραστηριότητες. Βεβαίως για το θέμα του προσωπικού ε, θα πρέπει πολύ σύντομα να έχουμε τα σχετικά ονόματα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Α, Σέντερ. Σας άκουσα τώρα να μας λέτε ότι στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό το Κοινοβούλιο θέλει πολύ, θέλει λίγο το Συμβούλιο και εσείς θα βρείτε τη μέση εδώ. Όμως το Ελληνικό Συνέδριο είπε και ξαναείπε ότι ένα από τα λάθη είναι το ότι έχουμε υπερβολικά φιλοδοξές πολιτικές και που δεν τις καλύπτουμε παρκώς από τον ε, προπολισμό. Είναι το βασικό στραβό που γίνεται. Και τώρα λέει η Επιτροπή ότι απαιτούνται από κράτη μέλη ε, περισσότερες πολιτικές για το προσφυγικό, μια άρτια πολιτική για άμυνα ε, και ασφάλεια με όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γύρω-γύρω. Οπότε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει κανείς, κάποιος δηλαδή που θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες για προτάσεις, από πλευράς Κομισιόν δηλαδή τι πρέπει να γίνει, αν τελικά να βρω τον προπολογισμό, τι είναι αυτό που θα κάνετε, είναι να ζητήσετε περισσότερα χρήματα για τον προπολογισμό, γιατί άνευ χρημάτων, άνευ πόρων, πολύ δύσκολα μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις πολιτικές. Δεν υπάρχουν πολιτικές χωρίς χρήμα. Ούτε ασφαλεία για άμυνα, ούτε πολιτική για το προσφυγικό. Ε, άρα, όμως, από θα βρουν τα λεφτά από την έρευνα, την απασχόληση, από τη Γεωργία. Μα γι' αυτό σας λέω, συνειδητοποιήστε ότι αν εσείς τελικά να λάβετε αυτό το χαρτοφυλάκι θα πρέπει να είστε ο πρώτος που θα πρέπει να ζητεί περισσότερα χρήματα. Όχι εμείς. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Εσείς όμως πρώτος θα πρέπει να βγείτε και να ζητήσετε περισσότερα χρήματα. Γι' αυτά όλα τα θέματα που συμφωνούν και τα τρία θεσμικά ότι είναι βασικά. Ε, γιατί δεν τι γίνεται, τι, κάνουν οι λαϊκιστές. Μα πάνε κόντρα. Άρα εσεί πρώτο να ζητήσετε περισσότερα χρήματα και εσεί θα πρέπει να ζητήσετε από πού θα βρεθούν αυτά. Η έκθεση μου ότι μα δίνει κάποιε ιδέε για τον προπολογισμό. Επίτροπε. Κύριε, Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, πιστέψτε ότι έχω και την βούληση και το θάρρος να το πράξω αυτό το τετραγωνισμό του κύκλου δεν θα το καταφέρουμε με τη δημοσιονομική πολιτική. Για το, για το δημοσιονομικό πλαίσιο, λοιπόν, σε σχέση με την ε, ιδιαίτερη μου πατρίδα, περιφέρειες οι οποίε χρειάζονται περισσότερα αντιθρωτικά μέσα. Στη συνέχεια ο εθνικό υπουργό, η τήρη της Γεωργίας, τη Οικονομία, του Πολιτισμού κτλ. Και όλα αυτά σημαίνουν το άθροισμα φιλοδοξιών που μας φτάνουν στο 150% των δυνατοτήτων μας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη σε μια πολιτική συνεκτική, σε μια πολιτική συνάγουσα των, ε, και συνάδουσα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ μέχρι το τέλος του έτους να έχω διατυπώσει προτάσεις οι οποίες θα σας πείσουν ότι είμαι σε θέση να δείξω και το θάρρος και την, τις ικανότητες που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Σβιευκά ένα λεπτό. Πρόεδρε, ξέρω ότι το θα έχετε κουραστεί, όμως εμείς από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σα υποβάλουμε τέσσερι ερωτήσει, συγκεκριμένε και σύντομες. Οπότε δεν θα καθυστερήσουμε την συζήτηση ιδιαίτερα. Είπαμε ε, ότι έχουμε το Brexit και την οικονομική του πλευρά που ε, είναι προφανές ότι έχει βαρύνουσα σημασία, οπότε εσείς έχετε αρμοδιότητα σε σχέση με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επιβιώσατε αυτό στην απάντησή σας ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει, να βοηθήσει τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από την Βρετανία. Εγώ θα σας ρωτήσω για το τι θα γίνει με αυτού που είναι ήδη συνταξιούχοι ή που θα γίνουν συνταξιούχοι στο άμεσο μέλλον, αυτοί που προέρχονται πάλι από την Μεγάλη Βρετανία, οι συντάξει θα καταβληθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Εσείς Πώ θα το χειριστείτε αυτό ω Επίτροπο Προπολογισμού, τι θα κάνετε στις συνομιλίε με του Βρετανού. θα πρέπει να συνεχίσουν να εισφέρουν οι Βρετανοί, θα πληρωθούν όλα μαζί, θα διαδεχθεί στην την υποχρέωση της Βρετανίας θα πει Βρετανία την ε, που καταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι οι συνταξιούχοι που είναι βρετανικής πικότητας έχει κατοχυρωμένα στα εκδοτικά δικαιώματα και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, κάποιος που είναι στο ενεργό δυναμικό, όπως είπε ο πρόεδρος, μετά το Brexit θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας από πλευράς εργατικών δικαιωμάτων, ώστε οι υπάλληλοι να μην υποστούν τις συνέπειες της αποχώρησης του, της χώρας ε, της οποίας την υπηκότητα έχουν προετοιμάζουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Η δική μου δουλειά είναι να ε, συλλέξω πληροφορίες για τα ποσά. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Και δυστυχώς Θα έχουμε λιγότερους ε, ε, υπαλλήλου από, την, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο στη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λιγότεροι είναι αυτοί που θα πληρώνουν και τις συντόξεις. Αλλά δεν αλλάζει αυτό τίποτα το, το Brexit δηλαδή σε σχέση με την καταβολή των συντάξεων θα πρέπει να γίνουν ομοδοποιημένες στατιστικές και να κάνουμε τον υπολογισμό. Τώρα, πώς θα γίνει αυτός ο υπολογισμός, νομίζω ε, ότι ως ε, εργοδότες ε, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε εμείς ε, τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των εργαζομένων και εσείς θα δώσετε την απαλλαγή όπως ήθιστε. Σίγουρα θα γνωρίζετε, Επίτροπε, ότι το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η πολιτική μας ομάδα αγωνίζονται για την σώτα ευκαιριών μεταξύ των δύο φίλων. Μα είπατε ότι σα ενδιαφέρει το θέμα και συμφωνεί με αυτή την πολιτική. Πετε μα συγκεκριμένα τι θα κάνετε τόσο ώστε να εξασφαλίσετε το ότι περισσότερε γυναίκε θα βρισκόνται σε διευθυντικέ θέσει ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν τη δημογραφική μεταβλητή που λέμε υπόψη τώρα με τις ε, ιδιωτικές εταιρείες τι γίνεται. Εσείς θέλετε να διαμεσολαβήσετε. Ε, στον διάλογο μας με το Συμβούλιο αλλά και για το τι θα γίνει σε σχέση με την ε, χώρα προελευσής σας για αυτή την υπόθεση, για αυτό το φάκελο Women on Boards. Οπότε τι θα κάνετε για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Ich glaube, zunächst rein. Ε, από πλευράς ε, συμβατικού και συνταγματικού δικαίου νομίζω υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εκπόνηση νομοθετικών πράξεων για την ενιαία αγορά πρέπει να ισχύει ισότητα των ευκαιριών, η απουσία της διακριτικής μεταχείρισης στα εργατικά δικαιώματα, η προστασία της σταδιοδρομίας. Δηλαδή, αντίθετα με αυτά που συμβαίνουν σε κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε ε, αρμοδιότητα να εκπονήσουμε νομοθετικές πράξεις. Στη Γερμανία υπάρχουν ε, σχετικές ε, διατάξεις για τα υποπτικά συμβούλια, αλλά όχι για τα διοικητικά συμβούλια ακόμη των επιχειρήσεων. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η επόμενη γερμανική κυβέρνηση και αν χρειάζεται να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, εμείς ε, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως πρότυπο. Θα λειτουργήσουμε εμείς μέτρα ως νόμονας για τους, υπολ... για τους υπολείπους. για τα ανώτατα στελέχη, για τους τμήματάρχες παραδείγματος χάρη, θα αποχωρήσουν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, θα συνταξιοδοτηθούν. Αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ούτω ώστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουμε την μελλοντική γενιά, κυρίως γυναίκε που έχουν την πλειοψηφία ω προ το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων. Θα πρέπει να τι ενθαρρύνουμε να υποβάλουν υποψηφιότητα για να καταλάβουν αυτέ τι χειρεύουσε θέσει. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Η επόμενη γενιά. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία κίνητρα, ε, επιμόρφωση των γυναικών, ενθάρρυνση των γυναικών ε, να αναλάβουν ηγετικές θέσεις. Ε, και στον ιστορικό κανονισμό η μόνη θετική διάκριση που υπάρχει είναι για τις υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειες ε, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε, ε, Επίτροπε. Έχουμε και άλλες δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι θέλετε να παραμείνει ελκυστικός εργοδότης Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα πετύχετε αυτό σας το στόχο συγκεκριμένα. Επίσης, προτίθεστε να αναθεωρήσετε τον ε, τρόπο προσλήψεων των υπαλλήλων από πλευράς ε, γεωγραφικού συντελεστή, γεωγραφικής μεταβλητής. Μας ενδιαφέρει αυτό ε, από πλευρά της ηχείας. Πώς η γεωγραφική ισορροπία, η δημογραφική ισορροπία θα αποτυπώνεται στις προσλήψεις θελκτικότητα του εργοδότη μετράται βάσει διαφόρων παραγόντων και μιλάμε για την αγορά εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ε, σύγκριση με την εθνική διοίκηση ή με την ε, βιομηχανία και είτε μιλάμε για διοικητικού υπαλλήλου, είτε ε, για μηχανικού, ε, για ειδικού ε, στον τομέα τη πληροφορική, για ειδικού στον ενεργειακό τομέα, προωθούνται οι νέοι. Και φυσικά είναι θέμα αποδοχών. Μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Επίσης, ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Ε, γιατί φτηνές δεν είναι αυτές οι δύο πόλεις. Ε, επίσης, επιδοτήσεις, ε, μέρημνα για τα παιδιά, ε, περίθαλψη, ε, η ποιότητα των ευρωπαϊκών σχολείων, ε, η προσφορά που έχουμε για την μετεκπαίδευση, οι ενδιαφέρουσες προσφορές για τους ε, υπαλλήλους ε, για τον χρόνο εργασίας 40 ε, ώρες αλλά θα ήταν λάθος να παρατείνουμε περαιτέρω αυτόν τον αριθμό ώρων εβδομαδιαίως θα πρέπει να κάνουμε ελκυστικές προσφορέ. όχι ε, απαραίτητα τις καλύτερες, αλλά γνωρίζοντας την κατάσταση των ανταγωνιστών μας. Ε, και πιστεύω ότι εξακολουθούμε να είμαστε ελκυστικοί εργοδότες ε, όταν ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Τώρα, όμως, Εάν μειώσουμε ή παγώσουμε για τόσα πολλά έτη τις αποδοχές ε, ή γραμμικά ε, μειώνουμε τον αριθμό των εργαζομένων και παρατείνουμε τον χρόνο εργασίας, ε, τι θα κάνουμε, θα, θα, σαν λεμονόκουπες θα τους απομυζήσουμε τους υπαλλήλους. Και ε, νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, θα είναι μετά ανταγωνιστικότερες οι εθνικές αγορές. Ε, μετά ε, είναι και το θέμα της επικότητας. Έχουμε τις βασικές 15 ε, υπηκότητες, είχαμε μέχρι στιγμής ε, που ήταν στο προσκήνιο. Ε, προσθέθηκαν οι νέες χώρες. Θα πρέπει Να δούμε επίσης ε, ποιοι αποχωρούν ε, στην ε, σύνταξη, δηλαδή να αυξηθούν από τις υπόλοιπες χώρες οι εργαζόμενοι και να καταλάβουν υψηλότερες θέσεις, ούτως ώστε να έχει ο υπάλληλο της νέας, του νέου κράτους μέλους προμελλοντικές προοπτικές στη σταδιοδρομία του. Ευχαριστούμε. Τελευταίος αλλά ο Πασκάλ Ντιγό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Οτίνγκερ, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή κατά την ε, ακρόση και επανειλημμένα μας είπατε ότι είστε πολιτικός ε, ε, έμπειρος. Οπότε θα πρέπει να αποκλείσουμε το σενάριο κατά το οποίο λέτε ότι να είναι ε, δημοσία σαν δηλώσεις και λέτε κάτι χωρίς να το σκεφτείτε. Όμως έχετε πει κάποια ομοφοβικά, κάποια ρατσιστικά πράγματα. Δεν, αυτά θα πρέπει να τα ανακαλέσετε. Εμείς ξέρουμε ότι θα ε, αναλάβετε τους ανθρώπινους πόρους. Δεν θέλουμε τώρα να ψάξουμε γιατί τα είπατε αυτά στο, ε, στις δηλώσεις σας. Και εγώ αν είμαι όμως ομοφιλόφιλος μπορώ να έρθω να εργαστώ για σας χωρίς να φοβηθώ ότι πρόκειται να υποστώ τις ε, συνέπειες. Δεν θα έπρεπε να το σκεφτείτε καλύτερα για να αποφύγετε τις δυσκολίες. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι βάδι Βιτεμβέργη σε πιο μεγάλη κλίμακα. Και περνάει δύσκολες ώρε η Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε να είσαστε πιο προσεκτικό και να ευχαριστήσετε τον Γεωργιούν και για την τιμή που σας έκανε. Αλλά να μην αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο των ανθρωπίνων πόρων. Ρίτα, εξέφρασα τη λύπη μου για αυτές τις ε, δηλώσεις. Και τα τελευταία 7 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω αποδείξει εμπράκτος ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιώ στο όργανο τη διακριτική μεταχείριση. Αν θέλετε ε, δείτε τις γενικές διευθύνσεις, στη DigiConnect, εκεί όπου ήμουνα, να δείτε πώς είναι η καμπύλη του προσωπικού. Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Ε, έχω επιτυχεί το στόχο μου. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να ανησυχείτε για την συνεργασία μαζί μου. Ε, δοκιμάστε με και ε, μπορείτε να περιμένετε από μένα ε, απουσία διακριτικής μεταχείρισης για την ε, καθημερινή δουλειά μου. Φτάσαμε στο τέλος της ανταλλαγής απόψεων με τις τρεις επιτροπές. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες για την προετοιμασία της ακρόασης. Οι συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού να, να παραμείνουν στην αίθουσα, συγγνώμη, Επιτροπής Προϋπολογισμού να παραμείνουν στην αίθουση, αίθουσα και στον τέταρτο όροφα να πάνε οι συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου των Οι συντονιστές της Επιτροπής ε, ε, Νομικών Υποθέσεων θα συνεδριάσουν αύριο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω και εγώ ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο που χαρέξει η κυρία Γεωργίευα στο ω προ τον έλεγχο των προπολογισμών. Ε, λύεται η συνεδρία και τώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ. Si vous le permettez, je voudrais indiquer. Αρτή. Από πλευρά του Προπολογισμού, θα σα πω ότι οι συντονιστέ θα συνδυάσουν σε αυτήν εδώ την αίθουσα και θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών σε πέντε λεπτά. Προβλέπετε όμως ένα λεπτό για τον κύριο Επίτροπο ούτω ώστε να διατυπώσει τα συμπεράσματά του. Έχετε το λόγο, Πίτροπε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους, για τις εκτιμήσεις τους. Σέβομαι όλες τις τοποθετήσεις, τις παίρνω όλες τα σοβαρά. Πολλές από τις ε, παρεμβάσεις δείχνουν ότι χρειάζεται να εμβαθύνουμε στις συνομιλίες μας με όλες τις ομάδες, τους ομιλητές, τους εντονιστές, τους εισηγητές και είμαι πεπισμένος βαθύτατα ότι έχουμε πληθώρα κοινών σημείων, πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε φέτος και στα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι μπορώ να δώσω την υπόσχεση πως θα ε, πάρει μεγαλύτερο χώρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις θέσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη Συνεδριάσεως, λέει ο κύριος Αρτουή. Οι συντονιστές παρακαλώ να μένουν στην αίθουσα.